Okay, colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Ανεξάρτητα από την συμμετοχή των συναδέλφων, πρέπει να συναντήσω τον Επίτροπο στις 4. Θέλετε να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, που το ξεκινήσουμε επισήμως. 25, 26, 27. Κάποιοι έχουν συνδεθεί χωρίς να έχουν πατήσει το κουμπί. Ένας ακόμα το πάτησε τώρα. Πολύ ωραία. Αυξάνει το αριθμός. Καταπληκτικά. Θα αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί, αν προκύψει. Ξεκινάμε λοιπόν με την συμβαστική τροπολογία α υπέρ. Κατά αποχές το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία υπαριθμών 5. εγκρίνεται 15 υπέρ, 13 κατά. Τροπολογία 6 υπέρ. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 7 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 8 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται Τροπολογία 9 και 10 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνονται, αλλά σε παληθεύσουμε ηλεκτρονικά για τις τροπολογίες 9 και 10 είναι ταυτόσιμες. Εγκρίνονται όντως 18 υπέρ, 11 κατά. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία Β δεν προβλέπεται χωριστή ψηφοφορία. Το σύνολο λοιπόν της συμβαστικής τροπολογίας Β ψηφίζουμε υπέρ. Μια μικρή σύγχυση βλέπω στην αίθουσα, λέει πρόεδρος. Βρισκόμαστε στη συμβαστική τροπολογία Β, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 24 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την τροπολογία 24 άρθρη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, όντως εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 26, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε για το σύνολο του κειμένου που τροποποιήθηκε, άρτη ψηφοφορία. Πέρας, 32 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε νομίζω τις ψηφοφορίες. Θα διακόψουμε την συνεδρίασή μας μέχρι τις 4 και 4, όπου προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Αλμούνια. Λυπάμαι που συνεχώς κάνουμε διακοπές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας αυτή την εβδομάδα. Αν μείνετε στην αίθουσα μπορώ να κάνω και τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και λίγο χρόνο λίγο αργότερα. Πρώτα απ' όλα, ενημέρωση για διαλόγους. Για την ύφη είχαμε στις 21 Νοεμβρίου τον ένατο γύρο συνομιλιών σημειώθηκε πρόοδος ε, για τη δομή της αγοράς, διαφάνεια προεμπορίας, ε, υποχρεώσεις G20, πρόσβαση σε υποδομές αγορών. Ο ε, επόμενος γύρος είναι τον Δεκέμβριο, μετά κεντρικά αποθετήρια είχαμε δύο τριλόγους τον Νοέμβριο, συζητήσαμε και κλείσαμε αρκετά πράγματα, πήγαν όλα στην τεχνική ομάδα ανοιχτά ζητήματα είναι οι κυρώσεις ε, για διακανονισμούς, ε, αντιμετώπιση των διακανονισμών, πτυχές του καθεστώτος τρίτης χώρας και το τι θα γίνει με τις τραπεζικές άδειες των αποθετηρίων. Επόμενη ε, συνεδρίαση 28 Νοεμβρίου Οδηγία λύσης ε, τραπεζών, ο 8 γύρος του διαλόγου ήταν στο Στρασβούργο που μας πέρασε, λύση χρηματοδότηση και εγγύηση καταθέσεων ήταν τα θέματα και επίσης όροι κρατικής παρέμβασης ε, και ως μια προληπτική ανακεφαλαιοποίηση αλλά και ως μέσο σταθεροποίηση σε συστημική κρίση. Επόμενος τριμερής διάλογος 27 Νοεμβρίου. Τρίψ. Ψηφίσαμε στην Ολομέλεια της προηγούμενης εβδομάδας και κατά πάγια τακτική η διαπραγματευτική ομάδα θα είναι ο εισηγητής και οι σκιώδης εισηγητές στην πολιτική συνεδρίαση για την εγγύηση καταθέσεων. Είχαμε την τέταρτη συνάντηση με τη Λιθουανική Προεδρία και την Κομισιόν 19 Νοεμβρίου με βάρος στο επίπεδο στόχου για το σχετικό ταμείο και το εάν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και υπό ποιους όρους όχι μόνο για καταθέσεις αλλά και σε διαδικασία έγκαιρης παρέμβασης ή λύσης. Σε σχέση με τα ταμεία μας, το Ταμείο Εγγύησης ε, ε Καταθέσεων έγινε Ταμείο Λύσης Τραπεζών και αντιστρόφως. Αναμένουμε επίσης περαιτέρω ενδείξεις για το τι θα γίνει σε αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα και ελπίζω να οριστικοποιηθούν σύντομα. Βεβαίως αυτό σχετίζεται με την οδηγία ανάκαμψης και λύσης τραπεζών. ζημίες ε, και αποζημιώσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα η διάσκεψη των Πρόεδρων έλαβε απόφαση για τις αρμοδιότητες. Το είπε νομίζω ο εισηγητής χτες, οπότε δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Αλλά η διάσκεψη των Προέδρων είπε πως ήταν επίγον να σημειωθεί πρόοδος και ειδικά να συμφωνηθεί ένα κοινό χρονοδιάγραμμα με την Γιούρη την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Πρέπει λοιπόν να ε, κινητοποιηθούν στην άλλη Επιτροπή. Λοιπόν, τα λέμε στις 4 ε, και 4. Ωραία, είμαι σίγουρο ότι ε, πολλοί είναι έξω. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν κάνουμε διάλειμμα γιατί διάφοροι φεύγουν έξω, τα μιλάνε στο τηλέφωνο, ξεχνιούνται μετά, βλέπουν άλλο κόσμο, συζητούν, τέλος πάντων. Επίτροπε Αλμούνια, καλωσορίσατε και πάλι στην Επιτροπή μας. Και πάντοτε κάνουμε πολύ καλές ανταλλαγές απόψεων. Ε, από τότε που έγινε η αρχική ακρόαση για να διοριστείτε, θα σας δώσω 10 <laughs> λεπτά και θα σας χρονομετρήσω. Και μετά θα περάσουμε στις ερωταπαντήσεις. Ε, και συλλογικά θα αφιερώσουμε ένα πεντάλεπτο για τις απαντήσεις ε, και αυτοί είναι οι κανόνες ε, και θα σας μουτρώσω αν ξεπεράσετε το χρόνο που σας αναλογεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που με καλέσατε και πάλι στην Επιτροπή σας. Ο συνήθως χαίρομαι που είμαι εδώ και μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Όταν προετοίμαζα την ομιλία μου και πλησιάζουμε και το τέλος του 2013, θεωρούσα σκόπιμο να κάνουμε έναν απολογισμό των δράσεών μας για το ολόκληρο το 2013 για να εξετάσουμε τα βασικά ζητήματα που θα εγκριθούν επίσης ε, κατά τη διάρκεια του 2014. Θα ήθελα να αφήσω με τα, αρχίσω με τα αντιτράς και τα καρτέλ. Το 2013 ασχοληθήκαμε με τους νέους ε, αναπτυσσόμενους ε, τομείς ε, κατά χρήση του συστήματος διπλώματων ευρεσιτεχνίας και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. για τα αντιτράστε η πρώτη έρευνα που έγινε στην βιομηχανία high-tech ήταν για την Google. Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε feedback από πάνω από 100 παίκτες της αγοράς για να έχουμε ένα βελτιωμένο set δεσμεύσεων από πλευρά τη Google. Ε, πρόσφατα εξήγησε εδώ στο Κοινοβούλιο με ποιο τρόπο εγώ προσεγγίζω αυτή την περίπλοκη έρευνα. Του προσεχεί μήνε ε, θα εξετάσουμε τα πορίσματα τη διαβούλευση και θα αποφασίσουμε ε, τι μέλη γενέστε για τι βασικέ αποφάσει που ελήφθησαν στον τομέα θα τονίσω πόσο σημαντικέ είναι οι δεσμεύσει τη Apple για του πέντε μεγαλύτερου εκδότε ηλεκτρονικών βιβλίων και την έρευνα που έγινε 561 ε, εκατομμύρια πρόστιμα για τη Microsoft γιατί δεν συμμορφώθηκε με ε, τα όσα είχαν αποφασιστεί το 2009. Πρώτη φορά επιβλήθηκε κύρωση σε εταιρεία ε, για αυτό το λόγο και το πρόστιμο δείχνει ότι πόσο σοβαρά παίρνουμε τη δέσμευση και την έμπρακτη συμμόρφωση. Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, για τα γενώσιμα φάρμακα και καθυστερημένη είσοδο στην αγορά επιβάλαμε 146 εκατομμύρια πρόστιμο στην Ρούμπε και άλλες εταιρείες. Επίσης έχουμε προϊούσες έρευνες ε, για ε, πρότυπα που σχετίζονται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ε, πρόκειται για οργανισμός πιστοποίησης, βιομηχανικής ε, πιστοποίησης για την διαλειτουργικότητα των συσκευών. Εκεί έχουν προχωρήσει περισσότερο οι έρευνες, σχετίζονται με τη Μοτορόλα, ενημερώσαμε την εταιρεία για τις ενστάσεις που έχουμε και μελετούμε τώρα την απάντησή τους. Η άλλη έρευνα σχετίζεται με τη Samsung που έχει αναλάβει δεσμεύσεις, ε, κάνουμε δοκιμές και αναλύουμε τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια, χρηματοπιστωτικές αγορές. Ε, πέρα από την εφαρμογή ε, του ειδικού καθεστώτος για τις τράπεζες, έχουμε προχωρήσει με τις έρευνες για το καρτέλε για τα... Ε, για το Λίμπορ και για τον Γιούριμπορ ε, και ε, κάνουμε νέες έρευνες για παρεμφερείς πρακτικές. Στείλαμε δήλωση ενστάσεων σε βασικούς, βασικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τα ασφάλιστρα κινδύνου και αντίστοιχες περιπτώσεις. Επίσης, κατάχρηση benchmarks σημειώθηκε και σε αγορές ισοτιμιών οι χρηματοπιστωτικές αγορές ε, πρέπει να είναι ασφαλείς ε, και διαφανείς ε, και ο κανονισμός συμμόρφωσης θα πρέπει να εφαρμοστεί. Μιλάμε για 146 εκατομμύρια πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε εταιρείε ηλεκτρονικών συστημάτων για τα αυτοκίνητα. Έρευνες γίνονται και για διάφορα άλλα τμήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Για τα καρτέλ, παραδείγματος χάρη, ασχοληθήκαμε με τα τσίπ για τα ευφύ αυτοκίνητα και ε, ε, προς το τέλος του έτους όμως κατέρευσαν όλες οι συνομιλίες ε, με όλους με όλε τι ε, αυτοκινητοβιομηχανίε. Συνεχίζουμε με τι δηλώσει ενστάσεων και θα ακολουθήσουμε τη συνήθεια διαδικασία. Για το Antitrust ε, έχουμε τι δεσμεύσει ε, τη Star Alliance, τη Air United και τη Air United, και τη Lufthansa. Συνεχίζουμε τι προσπάθειέ μα. Κάνουμε έλεγχο στην εταιρεία CES για τα ηλεκτρονικά κυκλώματα με την ε, Gazprom επίσης και για την ε, Ρουμανική ΔΕΗ. Επίσης 79 ε, εκατομμύρια πρόστιμα επιβλήθηκαν στην Πορτογαλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Διερευνούμε καταγγελίες για τη Σλοβακική, μια Σλοβακική εταιρεία τηλεπικοινωνιών επίσης. Ε, και επίσης ε, ε, ενδεχομένως έχουν υπάρξει παραβιάσεις για τη μεταφορά δεδομένων από άλλους φορείς της αγοράς. Θα ήθελα επίσης να σας εξηγήσω ότι έχουμε κάνει για τις συγχωνεύσεις και τους ελέγχους που κάνουμε. 219 καταγγελίες έχουμε λάβει σήμερα και 186 συμφωνίες τις έχουμε εγκρίνει χωρίς πρόβλημα. Στη συνέχεια έχουμε δεσμεύσεις και στις ε, στις 10 είμαστε στην πρώτη φάση και 10, ε, στις, στις υπόλοιπες 10 στη φάση 2. Για την UPS TNT ε, είναι η πρώτη έρευνα και για τη δεύτερη έρευνα Ryanair και Air Lingus και πέρα που δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ε, ήταν η περίπτωση της Intercontinental, παραδείγματο χάρη και την εξαγορά. Ε, ε επίσης, στην περίπτωση της Kabel Deutschland δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όπως είπα και νωρίτερα, ε, συνεχίσαμε τις εργασίες μας ε, με τις ε, τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, νέους κρατικούς ε, κανόνες ε, που τίθενται σε ισχύ από 1η Ογδόου. Ε, τους εξετάσαμε εν και της Τραπεζικής Ένωσης και ε, χάρη στην πραγματογνωμοσύνη που έχουμε αποκτήσει από την αρχή της ε, κρίσης, ε, κινηθήκαμε και τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε εξετάσει 68 αναδιαρθρώσεις τραπεζών και έχουν καθαριστεί 28. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα τέταρτο του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς στοιχείων ενεργητικού. Δεν έχει φυσικά ολοκληρωθεί το έργο μας. 25 περιπτώσεις εκκρεμούν, κυρίως στις χώρες προγράμματος, μνημονίου Ευρωζώνη. Το 2000, ε, από το 2008 μέχρι το 2012 εγκρίναμε ε, πολύ μεγάλα ποσά ε, κρατικών επιδοτήσεων που μόνο εν μέρει χρησιμοποιήθηκαν στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Μόνο ένα τρίτο των εγγυήσεων που είχε εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγήθηκαν από τα κράτη-μέλη τελικά. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, ε, η υποστήριξη κρατική προς το τραπεζικό σύστημα ως επιτοπλίστων πήρε την μορφή εγγύησεων και σχετικών μέτρων. Το 2012, 492 ε, δις κρατικών εγγύησεων είχαν εκταμιευθεί σε σχέση με το 1,6 δις, τρεις ε, συγγνώμη, ε, που ε, συνολικά εκταμιεύθηκαν το 2012 τα δύο δις χρησιμοποιήθηκαν όμως ουσιαστικά από αυτό το ποσό σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση 413 ε, δις ήταν το ποσό των ανακεφαλαιοποιήσεων και αυτό αντιστοιχεί στο 2,3% του ΑΕΠ ε, ολόκληρης της Ευρωζώνης το 2012 ε, με μέτρα κεφαλαιοποίηση υποστηρίχθηκαν τράπεζες σε 82 εκατομμύρια στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο Ιρλανδία 63 εκατομμύρια και στην Ισπανία 60. Royal Bank of Scotland 46 εκατομμύρια, 32 ε, δις, ε, ε, συγγνώμη, 22 δις η Μπάνκια και ούτω καθεξής. Για τους κρατικούς κανόνες θέλω να σας πω ότι τα κράτη-μέλη έχουν χορηγήσει όλα αυτά τα ποσά εγγυήσεων και 33 ε, δις έχουν λάβει ε, ε, σε τέλη εγγυήσεων τα κράτη-μέλη για το σύνολο των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί. Για το, στο τέλος του 2012 τα κράτη-μέλη πήραν 125 δις σε εισόδημα, σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη που προσέφεραν υπομορφή εγγυήσεων στις τράπεζες. Είχα εξηγήσει στην Επιτροπή την στρατηγική για τον εξυγχρονισμό εξυγχρονισμό των τραπεζών που ξεκίνησε το Μάιο του 2012. Ως προς το ρυθμιστικό σκέλος ε, του πακέτου έχουμε τον κανονισμό που εγκρίθηκε ε, το καλοκαίρι από το Συμβούλιο. Τι προβλέπεται ο Γενικός Κανονισμός για την βασική εξαίρεση και η εξαίρεση de minimis ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά θα εγκρίνει όλες αυτές τις εξαιρέσεις. Σε σχέση με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για το χρηματοπιστωτικό τομέα έχουμε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα που εγκρίθηκαν λίγο πριν την το 2012 οι νέε περιφερειακέ κατευθυντήριες γραμμέ εγκρίθηκαν πέρσι τον Ιούνιο και ε, για τι τηλεπικοινωνίε ε, αυτό έγινε πριν από δύο εβδομάδε. Οι περιφερειακές κατευθυντήριε γραμμέ ε, θα δώσουν του κανόνε για τα ΜΜΕ και θα εγκριθούν στι αρχέ του Ιανουαρίου. Θα συνεχίσουμε με την αεροπορία, του κανόνε για τι μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες, για την έρευνα και την καινοτομία και στη συνέχεια τις περιβαλλοντικές κατευθυντήριες αυτό σημαίνει ότι τα βασικά στοιχεία του πακέτου εξυγχρονισμού ε, θα πρέπει να υπάρχουν κατά το πρώτο ήμιση το 2014 και θα αρχίσουν να ισχύουν από 1η ε, Εβδόμου το 2014 το αργότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, ανεκτήμητη βοήθεια του ε, βελτιώσατε το, ε, τη διατύπωση της ε, νομοθεσίας. Στη συνέχεια, οι κυρώσεις για αντιτράστε που ενέκρινε τον Ιόνιο το Ευρω... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προδέψει ήδη το κείμενο στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο ε, Ανταγωνιστικότητα. ελπίζουμε θα υιοθετήσει την ίδια γραμμή για το Κοινοβούλιο. όπω ξέρετε έχει εγκριθεί μια γραμμή από τη δική σα Επιτροπή και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για το έγγραφο εργασία. Ε, σημειώνουμε ότι το Κοινοβούλιο επίση έχει εκφράσει την ισχυρή επιθυμία του να ολοκληρωθεί πριν εκπνεύσει η θητεία αυτό το νομοθετικό πακέτο για το αντιτράστε, τους κανόνες αντιτράστε, Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε ανεξαρτήτως από την καθυστέρηση που σημειώνουμε σημειώνεται στις και στι δύο επιτροπές. Εάν τελικά τα καταφέρετε προτού λήξει η θητεία, νομίζω όλοι όσοι είναι ε, να λάβουν αποζημιώσεις, ε, αν δεν τα καταφέρουμε θα λάβουν ένα πάρα πολύ ε, αρνητικό μήνυμα. Τώρα η πρωτοβουλία για την αυλούστευση των συγχωνεύσεων πάρα πολύ σημαντικό για τις εταιρείε και θα συντομεύσω και την ομιλία μου παρότι ε, βλέπω ότι μάλλον θα ξεπεράσω τα 10 λεπτά. Ε, για το 2014 προτεραιότητα είναι η αναθεώρηση για τους κανόνες αντιτράστε για τον κανονισμό των μαζικών εξαιρέσεων για τις μεταφορές στις τηλεπικοινωνίες. Επίσης η νέα οδηγία για τις πληρωμές, ε, κυρίως ο κανονισμός ε, για τα τέλη θα εργαστούμε σκληρά ούτως ώστε να διευκολύνουμε τη διαδικασία συναπόφασης και για τα δύο ζητήματα και ε, ε, ποιες είναι οι εξελίξεις της διεθνής μας σχέσης την περασμένη εβδομάδα. Ε, Memorandum of Understanding ε, γράφει στην Ινδία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ε, MOUs ε, με τέσσερι από τις πέντε BRICS και σκοπεύουμε το, την επόμενη, το επόμενο μνημόνιο συμφωνίας να το διαπραγματευτούμε με την Νότιο Αφρική δεύτερης γενιάς συμφωνία υπέγραψε η Ελβετική, Ομοσπονδία, ε, η Ελβετική Ομοσπονδία και στην ε, ε, οι συζητήσεις αναμένεται να αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα ένα ε, κάτι άλλο ενδιαφέρον επίσης για τον ανταγωνισμό είναι η TTIP, ε, η Νέα Διατλαντική Εταιρική Σχέση για τις Επενδύσεις. Ε, θα καλύψουμε τα αντιτράστα, τους κανόνες αντιτράστα, τις συγχωνεύσεις, τις εταιρείες κρατικής ιδιοκτησίας, τις κρατικές επιδοτήσεις και ευελπιστούμε να έχουμε μια ευτυχή εξέλιξη γενικότερα για τις διαπραγματεύσεις TTIP και σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Σε ευχαριστώ. Περνάμε τώρα κατευθείαν στις ερωτήσεις. Ε, ο Πάμπλο για το ΕΛΚ. Ε, ευχαριστώ, Σάρων. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ, κύριε Επίτροπε, σε ένα ζήτημα το οποίο θέσατε στο τέλος της ε, ομιλίας σας. Η έκθεση μύφη για... με συγχωρείτε, για τα τέλη τα πολυμερή των συναλλαγών. αν ξέρετε τι θα συμβεί. Φοβάμαι πώς θα δημιουργήσουν ε, ένα αποτέλεσμα αντίθετο από αυτό το οποίο επιθυμούμε. Επίσης, η αξιολόγηση αντικτύπου δεν έχει λάβει υπόψη όλα αυτά τα ζητήματα, ειδικά όταν μιλάμε στο τι επίδραση θα μπορούσαν να έχουν σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα που υπάρχουν στην Ευρωζώνη. Επίσης ε, μπορεί να υπάρξει ένα πλαφόν σε μια αγορά όπου υπάρχει μεγάλη χρήση πιστοτικών καρτών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλη αγορά με μικρότερη χρήση πιστοτικών καρτών. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες διαφορές. Θα ήταν χρήσιμο να μας δώσετε κάποιες ε, περισσότερες ε, πληροφορίες. Έχει διατηρηθεί αυτή τη στιγμή η ιδέα των πλαφών γιατί δεν θέλουμε να αφαιρούμε πράγματα αλλά θέλουμε κάποια διαβεβαίωση από εσά για να είμαστε σίγουροι ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ βεβαίως να έρθω στο κοινοβούλιο να σας μιλήσω για τις λεπτομέρειες του ζητήματος αυτού. Μοιάζει περίπλοκο, αλλά είναι απλό. Στην πράξη. Έχουμε την ιδέα της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, κάτι το οποίο σημαίνει πως ε, οι μεγάλοι παίκτες ε, στις πιστοτικές και χρεωστικές κάρτες θα έχουν ένα σημαντικότερο ρόλο και αν είναι να χρεώνει κανείς τους πελάτες για τη χρήση κάρτας αντί για τη χρήση μετρητών υπάρχει ένα εναλλακτικό κόστος το οποίο μπορεί να καλυφθεί από τις εταιρείες των καρτών. Μπορούν να ωφεληθούν από αυτό γιατί ωφελούνται από τη μείωση του κόστους χρήσης μετρητών. Και λόγω των επενδύσεων που έχουν γίνει, όχι με βάση τον προτινόμενο κανονισμό, αλλά πριν από την πρόταση, όσον αφορά τις υποθέσεις ανταγωνισμού, μία αφορούσε τη Mastercard, μία άλλη τη Visa, ε, ξέρουμε πως ε, αυτό είναι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε για να μην υπάρξει κατάχρηση ε, τη της ε, θέση σε μια αγορά όπου δεν υπάρχει διαφάνεια γιατί οι καταναλωτές δεν ξέρουν ποτέ ε, ποια είναι τα τέλη που χρεώνει η εταιρεία της πιστοτικής κάρτας και συχνά δεν ξέρουν πως οι ε, λιανοπολιτές προσπαθούν να τους φορτώσουν αυτά τα έξοδα. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση γιατί έγινε μια έρευνα για τη λειτουργία του ανταγωνισμού. Είδαμε τι έγινε στη ΣΥΠΑ όπου δράσεις εκ των υστέρων δεν είναι τόσο αποτελεσματικές και αυτό ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις και οπωσδήποτε σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό θεωρούμε πως ο κανονισμός είναι πολύ πιο αποτελεσματικός και με τον Επιτρόπο Παρνιέ το Σώμα των Επιτρόπων ε, κατέληξε σε αυτή την πρόταση κανονισμού που υπέβαλε στο Κοινοβούλιο, αλλά γεγονό είναι πως είναι περίπλοκες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ να ξαναέρθω και να σας ε, ξαναμιλήσω για να εξηγήσω το γιατί θεωρούμε πως είναι σωστός αυτός ο κανονισμός και ποιο θα έπρεπε να είναι το επίπεδο των πλαφών, ε, όπως παρουσιάζεται στην πρόταση. Σας ευχαριστώ. Ελίζα Φεραίρα για τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σε σχέση με το Asset Quality Review που θα γίνει για τις ευρωπαϊκές ε, τράπεζες ε, προτού αρχίσει να ισχύει ο ενιαίος μηχανισμός υποπτίας. Κατά τη γνώμη σας, Ποιο θα είναι το βάση του ρυθμιστικού πλαισίου η ερμηνεία που θα κάνετε των κανόνων ανταγωνισμού. Τι εννοώ. Θα ζητήσετε μια συγκεκριμένη τιμή από τους βασικούς μετόχους και από τους junior μετόχους ε, ανάλογα με τη θέση που έχει αυτή η συγκεκριμένη τράπεζα ε, στη συγκεκριμένη χώρα η δυνατότητα παρέμβασης ε, των κρατών ε, πιστεύετε ότι θα οδηγήσει σε ανισορροπίες προτού αρχίσει να ε, ισχύει ο κανονισμός για την ενιαία Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή ο ESM θα μπορέσει να κάνει άμεσες ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών. Αυτή είναι μια άλλη ερώτηση. Ε, εφόσον επιδιώκουμε ε, να δημιουργήσουμε μια πραγματική ε, τραπεζική ένωση, θα αφήσουμε ένα διακυβερνητικό μηχανισμό να αποφασίσει για ανακεφαλαιοποιήσεις και στήριξη τραπεζών σε διάφορες χώρες, γιατί μπορεί να ανακύψει μια πάρα πολύ περίπλοκη κατάσταση ως προς την άνηση με μεταχείριση και τις τρευλώσεις ανταγωνισμού. Θα ήθελα παρακαλώ να τοποθετηθείτε και για τα δύο ζητήματα. Σας ευχαριστώ κυρία Φερέιρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συγκεκριμένα ο Μάριο Ντράγκη, και ήρθε και σας μίλησε, αν δεν κάνω λάθος, για το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Προτού αρχίσει να ισχύει ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να κάνει μια σφαιρική ανάλυση προκειμένου να δει την κατάσταση υγείας του τραπεζικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως για τις τράπεζες εκείνες οι οποίες θα ταχθούν στην ανάλυση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναφέρομαι σε 130 περίπου ευρωπαϊκές τράπεζες. Τώρα, όσον αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, το Asset Quality Review, αυτό θα είναι ο πρώτος μας στόχος και δεύτερος στόχος θα είναι τα stress tests. Οι δοκιμές αυτές αντοχής που θα γίνουν για ορισμένε τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για τις δύο λοιπόν αυτές δράσεις, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προσπαθήσει να δει πώς συμμορφώνονται οι ευρωπαϊκές τράπεζες με τις απαιτήσει κεφαλαϊκών με τι κεφαλαικέ απαιτήσει και του σχετικού κανόνε θέλουν να δουν ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν οι τράπεζε, και αν οι τράπεζες ανταποκρίνονται στου συγκεκριμένου κανόνε που έχουμε πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα τα stress tests αυτά καθ' αυτά, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δει σε ποιο βαθμό ενδεχομένω να επιδεινωθεί η κατάσταση για ορισμένε ευρωπαϊκέ τράπεζε. Και για αυτή την κατηγορία των τραπεζών η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να δει πώ θα ανταπεξέλθουν οι τράπεζε αυτέ. Αν δηλαδή υπάρχουν κάποιες τράπεζες οι οποίες δεν τα βγάλουν πέρα, δεν καταφέρουν να έχουν θετικά αποτελέσματα στα stress tests, τότε η ενιαία αρχή επιτήρησης θα πάρει μια απόφαση εκ νέου ανακεφαλοποίησης των τραπεζών αυτών, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε αρνητικό σενάριο ή ώστε να καταφέρουμε τουλάχιστον να διαχειριστούμε ένα οποιοδήποτε αρνητικό σενάριο. Όσον αφορά λοιπόν τις κατευθυντήριες γραμμές που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων προς τον τραπεζικό τομέα και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αυτό είναι κάτι που θα μας πασχολήσει όλος ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια του 2014. Σε περίπτωση εξυγίανσης εκαθάρισης τράπεζας ή ανακεφαλοποίησης τράπεζας, τότε η εν λόγω τράπεζα θα υπόκειται στην εξή διαδικασία. Ενδεχομένως να κρυθεί ότι χρειάζεται λοιπόν επιπλέον κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης. Θα πρέπει επίσης να γίνει μια αναθεώρηση και αξιολόγηση της κρατικής ενίσχυσης που δίδεται προς την τράπεζα αυτή και να δούμε στη συνέχεια αν αυτό συνάδει με το σχέδιο μεταρρύθμισης αναδιοάρθρωσης το οποίο θα έχει υποβάλει εκ των προτέρων η ίδια η τράπεζα. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα καταστήσει εκ νέου την τράπεζα βιώσιμη και ότι θα καταφέρει να λειτουργήσει ομαλά στην αγορά η τράπεζα αυτή χωρίς να χρειαστεί στο μέλλον περαιτέρω ανακεφαλοποίηση, τότε η λόγω τράπεζα θα πρέπει να καλύψει μόνη της τις κεφαλαιοκές απαιτήσεις της και προτού δοθεί άδεια για κρατική ενίσχυση προς την τράπεζα αυτή, θα πρέπει να γίνει μια διαβούλευση με τους μετόχους θα πρέπει να εξετάσουμε τον ισολογισμό της τράπεζας αυτής, να δούμε ότι υπάρχουν όντως οι απαραίτητοι πόροι. Θα πρέπει επίσης να δούμε ποια είναι τα υβριδικά προϊόντα τα οποία διαθέτει η τράπεζα αυτή, να εξετάσουμε καλύτερα το ενεργητικό και το παθητικό του ισολογισμού της και θα πρέπει να δούμε επίσης πώς θα καταφέρουν να συμβάλλουν οι λεγόμενοι junior μέτοχοι. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε πιστεύω να καλύψουμε τις κεφαλαικές απαιτήσει που θα έχει αποφασίσει ο... η ενιαία αρχή ελέγχου, η ενιαία αρχή εποπτείας. Μόνο αφού ικανοποιηθούν όλα τα κριτήρια αυτά, θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγκριση για κρατική ενίσχυση προς την τράπεζα αυτή. Όπως σας είπα όμως θα πρέπει πρώτα να γίνει μια διαβούλευση με τους μετόχους, με τους junior μετόχους και τότε μόνο ενδεχομένως να εγκριθεί μια κρατική ενίσχυση για την τράπεζα αυτή, μια πολυμερής ενίσχυση, όπως είδαμε στην περίπτωση της Ισπανικής Τράπεζας, όπου χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ESM, προκειμένου να δοθούν κάποια κεφάλαια όχι μόνο από τον κρατικό κλάδο, αλλά και από τον ιδιωτικό κλάδο. Όμως το σύστημα αυτό λειτουργήσε προτού εγκριθεί το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτού δηλαδή δημιουργήσουμε, προτού θεσπίσουμε το σύστημα του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας. Νομίζω ότι το σύστημα αυτό το οποίο σα προτείνουμε είναι θετικό. Έχω εξετάσει κάπω τα αριθμητικά δεδομένα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και τους σχετικούς κινδύνους για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους κίνδυνοι δηλαδή που απορρέουν από μια περαιτέρω διάσωση του τραπεζικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που είδαμε είναι ότι 60 περίπου τράπεζες εντάσσονται στα προγράμματα αυτά, θα μπορούσαν δηλαδή να ενισχυθούν κρατικά. Ξέρετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν πλέον να καλύπτουν με δικά τους χρήματα την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν στο μέλλον οι τράπεζες να μπορούν να καλύψουν από μόνες τους τις ανάγκες κεφαλαιοποίησής τους. Ξέρετε ότι μέχρι στιγμής ήταν οι φορολογούμενοι αυτοί οι οποίοι διέσωσαν κυρίως τις τράπεζες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απόλυτα λογικό, δίκαιο και πολιτικά ευκταίο να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή που σας περιέγραψα. Θα περιέχεται μάλιστα σε όλο σύστημα μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση εκείνη όπου θα πρέπει να γίνει μια ιεράρχηση του ποιος θα πρέπει να συμβάλλει στην διάσωση των τραπεζών, θα πρέπει να αξιολογηθούν όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι. Πάντως, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, από όσο γνωρίζω, εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρησιμοποιούμε κυρίως συστημικά μοντέλα τραπεζών, τα οποία δεν είναι καθόλου συστημικά στην ουσία. Μπορείτε στη συνέχεια να μου απαντήσετε για ε, το ESM. A contestarle. Pero... Ε. Ζητήστε από τον πρόεδρο του Eurogroup να σας απαντήσει. Forma parte de eh, decisiones, las toman Πρόκειται για ένα διακυβερνητικό σύστημα. Ε, λαμβάνονται οι αποφάσεις από τα κράτη-μέλη. Σας είπα ότι στην περίπτωση της Ισπανίας με την εφαρμογή της ε, συμφωνίας από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 ο ESM έδωσε κεφάλαια στην Ισπανία για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και αυτό θεωρήθηκε κρατική ε, χορήγηση, κρατική επιδότηση. Αυτό όμως ε, επηρεάζει τις ε, αγορές και δημιουργούνται ε, στρεβλώσεις ανταγωνισμού. Έτσι, ποια κριτήρια εφαρμόζονται. πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα βασικό στοιχείο στο σχέδιο της Τραπεζικής Ένωσης που ευελπιστώ ότι θα λάβει σάρκα και ωστά το ταχύτερο δυνατόν. Πρέπει λοιπόν να σπάσουμε τα δεσμά ανάμεσα στο δημόσιο χρέος και τον ισολογισμό των τραπεζών. Ε, το αντίθετο συμβαίνει ουσιαστικά. Ε, ε, εστιάζουμε τι προσπάθειέ μα στι χώρε που αντιμετωπίζουν και του μεγαλύτερου κινδύνου. Πρόεδρο, ναι, αλλά τελικά τα κεφάλαια είτε είναι στον ESM είτε προέρχονται από κάπου αλλού. Είναι από τον δημόσιο κορβανά. Οπότε κατά τη διαστολή με τα κεφάλαια των τραπεζών. Ε, ξαναλέω ότι η βάση του άρθρου 107 ε, είναι πόροι των κρατών μελών. Απάντηση. Ναι, εκτός και αν οι πόροι προέρχονται από τον ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούνται ως κρατικά ποσά και άρα εξετάζονται βάσει των κανόνων για τις κρατικές επιδοτήσεις. Και δεν υπάρχει επιλεξιμότητα, δηλαδή υπάρχουν κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρήση αυτών των κονδυλίων δεν εκφεύγουν ε, του ελέγχου εκτός αν έρχονται από τον προϋπολογισμό. Ε, πρόεδρος ε, και ε, εξισώνονται έτσι αυτοί που είναι εντός και αυτοί που είναι εκτός της Ευρωζώνης όμως με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων για τους... Ε, στο Σάρων κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Θυμάμαι και την προηγούμενη φορά που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον Ανδρέας Σουάμπ ήρθατε στην διάσκεψη που είχαμε κάνει για την ε, περίπτωση της ε, Google. Ίσως λοιπόν ο Ανδρέας να έχει κάποια σχετική ερώτηση. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα επιτόκια. Τα τελευταία νούμερα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Σεπτεμβρίου μας είπαν πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ζητάνε δάνεια κάτω από ένα εκατομμύριο ευρώ, οι περισσότερες δηλαδή πληρώνουν 2,7% επιτόκιο παραπάνω από τις εταιρείε που ζητάνε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ δάνειο. Εγώ είμαι Καταλανός, ξέρετε πως έχουμε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό το ερώτημα προκύπτει πάντα. Έχουμε λοιπόν ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας εδώ πέρα, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θέλουν να μάθουν το τι θα κάνει η Κομισιόν για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τρεμόσα. Πρώτα απ' όλα μια διευκρίνηση. Με μεγάλη χαρά συμμετείχα στην ημερίδα που συνδιοργανώσατε με τον Ανδρέας Σουάβα, αλλά δεν είπα πως έχει υπάρξει κάποια συμφωνία επί της αρχής με την Google. Η Google έκανε κάποιες προτάσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή αναλύουμε. Δεν μίλησα για συμφωνία επί της αρχής. Τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναι βεβαίως είναι σαφές πως αν μιλήσουμε ειδικά για την Ευρωζώνη υπάρχουν ε, διαφορετικές συνθήκες ε, που ισχύουν ε, για την λήψη δανείων ειδικά από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στις κεφάλαια αγορές και η δυσκολία αυτή στην πρόσβαση οφείλεται σε διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα σχετίζεται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την σταθερότητά τους. Αυτά τα ιδρύματα όμως διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Δηλαδή αν υπάρχει ένα κομμάτι του τραπεζικού συστήματος υπό αναδιάρθρωση ή αν στην ίδια χώρα το τραπεζικό σύστημα έχει δυσκολίες ή πρέπει να ενισχύσει τα κεφάλαιά του για να αντιμετωπίσει τις ε, καθυστερούμενες πληρωμές κτλ. Τότε προφανώς ε, οι πόροι που έχουν οι τράπεζες για να δανείσουν ε, είναι λιγότεροι. Το δεύτερον αφορά το κόστος του χρήματος για τις τράπεζες. Κάποιοι από αυτούς τους πόρους, ειδικά όταν μιλάμε για τράπεζες που εστιάζουν σε δάνεια προς μικρόμεσες επιχειρήσεις, είναι οι καταθέσεις κατοπισμένοι πως δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλο κόστος παρά το ότι σε κάποιους τομείς υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά για κάποια πιστοτικά ιδρύματα υπάρχει ανάγκη να προσφύγουν στις ε, χρηματαγορές. Και εδώ πέρα πάλι διαφέρουν τα επιτόκια γιατί δεν βασίζονται ε, απαραίτητος ε, στη φερεγγιότητα του πιστοτικού ιδρύματος, αλλά το παραπάνω κόστος που οφείλεται στη χώρα όπου εδρεύουν. Έτσι. Ξέρω βεβαίω πως τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ από το καλοκαίρι του 2012. Αυτό το έξτρα κόστος του κινδύνου χώρας έχει πέσει κατά πολύ αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν σημαντικές ε, διαφορές όσον αφορά το κόστος ε, της ε, πίστης και βέβαια πρέπει να δούμε και τις δυσκολίες και γενικά το ότι μειώνεται η ροή της πίστης και πρέπει να λάβουμε υπόψη βεβαίως και τη ζήτηση, όχι μόνο την προσφορά. Αν δούμε τη ζήτηση σε χώρες όπου υπάρχουν πολλές χρεοκοπίες και υψηλό επίπεδο χρεών και υπάρχει και μηδενική ανάπτυξη και η ζήτηση για δάνεια θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Οπότε δεν υπάρχει κίνητρο από πλευρά φερικαιότητας να κάνουν κάτι οι τράπεζε γιατί μπορεί να έχουν κάποιο περιθώριο να δώσουν δάνεια αλλά αντιμετωπίζουν ε, κινδύνους από πλευράς αυτών που ζητούν τα δάνεια. Οπότε και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τώρα. Προφανώς, αν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα κοιτάνε την ε, προσφορά αντί για τη ζήτηση. Και αν είσαι τράπεζα, το βλέπεις αντίστροφα. Οπότε είναι ανάλογα με το ε, σε ποιον μιλάει κανείς. Βεβαίως ε, πρέπει να υπάρχει ισορροπία και στις δύο πλευρές της αγοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βίκη τώρα για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τα τελευταία χρόνια είχατε πάρα πολύ δουλειά. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί θεωρούμε πως η πολιτική ανταγωνισμού είναι πάρα πολύ σημαντική για να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και έχω διάφορες ερωτήσεις που θα ήθελα να κάνω και χαίρομαι που θα απαντήσετε και μετά τη συνεδρίαση. Τώρα, για ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό αφορά την επόμενη γενιά πυρηνικής ε, ενέργειας. Πρέπει δηλαδή ε, να παίξετε τον ρόλο σας, να υπάρχουν ε, επενδυτές και οι επενδυτές σε κάθε είδος ενέργειας να έχουν μια βεβαιότητα για τις αποφάσεις που θα λάβουν. Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν. Μπορείτε μήπως να με διαβεβαιώσετε πως οι αποφάσεις που θα λάβετε ε, θα βασίζονται σε ίσους όρους ανταγωνισμού, θα αντικατοπτρίζουν το ότι τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν το δικό τους ενεργειακό μείγμα και επίσης ότι θα είναι τεχνολογικά ουδέτερες, οπότε δεν θα υπάρχει παρέμβαση ε, και θα λέμε αυτή η τεχνολογία μας αρέσει και η άλλη όχι. Προφανώς ε, ερχόμαστε σε μια περίοδο αλλαγής της Κομισιόν. θεωρείτε ότι το θέμα αυτό θα περάσει στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ θα δυσφαλίσουμε θα έχετε όλες τις πληροφορίες στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Καθώς προετοιμάζουμε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον, ε, η υπερνική ενέργεια είναι στο κέντρο συζητήσεων, συναισθημάτων κτλ. Και εγώ προσπαθώ πάντα να κάνω μια ανάλυση ψυχρή, ήρεμη και όσο δυνατόν πιο λογική και προσπαθώ να κρύψω τις δικές μου ε, προτιμήσεις, το δικό μου ενεργειακό μείγμα. Έχω κάποιο, αλλά βεβαίως ως ε, αρμόδιος ε, για τα θέματα αυτά πρέπει να σεβαστώ την συνθήκη που λέει πως κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει το τι θα κάνει όσον αφορά το τι ενέργεια θέλει να χρησιμοποιήσει και γι' αυτό το λόγο όταν υπέβαλα στις υπηρεσίες της Κομισιόν, έτσι, όχι σε δημόσια διαβούλευση, στις διάφορες γενικές διευθύνσεις. Το πρώτο σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών ενέργειας και περιβάλλοντος ζήτησα να μπει εντός παρενθέσεων στην περίπτωση που αποφασιστεί πως τα κριτήρια αξιολόγησης μιας επένδυσης σε πυρηνική ενέργεια θα έρθουν στο γραφείο μου, ποια θα είναι αυτά. Δηλαδή γράψτε τα κριτήρια εκ των προτέρων ε, για να αποφύγουμε τις συναισθηματικές συζητήσεις, τις εντάσεις κτλ. Και να πούμε ομά σε όλους πώς η Κομισιόν θα αξιολογήσει κατά περίπτωση μια πιθανή πρόταση για επένδυση σε πυρηνική ενέργεια, χρησιμοποιώντας τη συνθήκη και μόνο αυτήν. Δεδομένων των συζητήσεων και της παρερμηνίας ε, των προθέσεών μου, που ήταν να έχουμε μια λογική συζήτηση, ζήτησα από τους συναδέλφους μου σε μια συνάντηση στο Στρασβούργο το Σεπτέμβριο να μου επιτρέψουν να διαγράψω τη λέξη ε, πυρηνική ενέργεια από τις κατευθυντήριες γραμμές γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως θα λάβω, πως και έγινε, μία πρόταση που θα υπονοεί πως υπάρχουν σοβαρές ε, αμφιβολίες για την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων. Ας αξιολογήσουμε αυτή την πρόταση και τις άλλες ε, μόνο με τη συνθήκη. Και αυτό συμβαίνει. Οπότε, σεβασμό για τις αρμοδιότητες και τα προνόμια των κρατών μελών, μόνο αυτά μπορούν να αποφασίσουν επί τόπου τι πηγές ενέργεια θα χρησιμοποιηθούν. Δεύτερον, η ενέργεια αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς ε, στήριξη του, της κοινής γνώμης, γιατί βεβαίως οι εξωτερικότητες ε, της φαινικής ενέργειας είναι μεγαλύτερες από αυτές ε, των ε, ανεμογεννητριών και της ηλιακής ενέργειας, αλλά ας το δούμε από την αρχή με βάση τη συνθήκη. Έλαβα μία πρόταση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, Ξέρουμε πως κάποια άλλα κράτη-μέλη εξετάζουν παρόμοια προγράμματα. Οπότε δεσμεύομαι πως όταν έχουμε μια θέση η ανάλυση θα είναι ήρεμη, εις βάθος, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα οποία θέλει το κράτος μέλος που έχει προτείνει κάτι, αλλά και τις διάφορες απόψεις εντός της Κομισιόν και όλων των εμπλεκομένων μέρων πριν προτείνω ή μάλλον προτείνει ο διάδοχός μου τις ε, συναδέλφους της ε, κάποια απόφαση. Δεν ξέρω πότε. Σας ευχαριστώ για τους πράσινους ο Φιλίπ Λαμπέρτς. Σας έκλεψαν την ερώτηση με την πυρνική ενέργεια. Όχι, όχι. Αλλά είναι ενδιαφέρον ε, η δίκη που είναι υπέρ της αγοράς να υπερασπίζεται μια ενέργεια η οποία δεν είναι βιώσιμο χωρίς κρατική στήριξη. Απλά είναι διασκεδαστικό Βίκυ γιατί είσαι υπέρ της αγοράς όταν σε βολεύει αλλά όχι τόσο όταν δεν σε βολεύει. Ε, τέλος πάντων. Κύριε Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να έχω τα αριθμητικά αυτά δεδομένα τα οποία αναφέρατε στην αρχική σας δήλωση. Θα ήθελα επίσης όμως να γνωρίσω και ποια είναι η αποψή σας όσον αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε νέα διάσωση των τραπεζών, ιδίως στα πλαίσια της Νέας Τραπεζικής Ένωσης. Από τη μια έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για το τραπεζικό τομέα. Είναι πολύ θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια σχετική ανακοίνωση. Πρέπει να εφαρμοστούν τώρα όμως οι γραμμές αυτές οι κατευθυντήριες. Στα πλαίσια της ε, οδηγίας Μπέρτιν, οποία διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή, ως ποιο βαθμό μπορούμε να εφαρμόζουμε το bail-in και υπάρχει δυνατότητα bail-out ως ίστατη λύση τελικά, έσχατη λύση, αν τελικά τεθεί εν κινδύνο η ίδια η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όμω γιατί ενδεχομένω να χρησιμοποιήσουμε πολύ εύκολα τη χρηματοπιστωτική αστάθεια ω πρόσχημα για να διασώσουμε εκ νέου τράπεζε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έναν δικαστή που θα έχει ένα ρόλο διαιτητή και ο οποίο τελικά θα κρίνει πότε μπορούμε τελικά να περάσουμε από ένα καθεστώς bail-in σε ένα καθεστώς bail-out ή αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ποσοστό bailout αφού έχει εφαρμοστεί πρώτα μια λύση bail-in. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει αυτό τον διτητικό ρόλο. Αν πρέπει τελικά να αποφευχθεί όντω μια πολύ μεγάλη χρηματοπιστωτική καταστροφή και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα βαθμό bailout, θα ήθελα τότε ένα υπεύθυνο υψηλόβαθμο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μια σχετική άδεια για κάτι τέτοιο. Αν όμω τότε έχουμε πραγματικό πρόβλημα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αν εξεκριβωθεί δηλαδή κάτι τέτοιο και αν έχουμε τελικά κρατικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες, θα πρέπει αυτές να συνάδουν με τους κανόνες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να ξέρουμε και ποιες διορθωτικές δράσεις μπορούν να ληφθούν. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι έχουμε δύο αποφάσεις οι οποίες θα υποβληθούν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια θα είναι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Η Γενική Διεύθυνση η Μάρκτα είναι αυτή η οποία θα κρίνει αν τελικά τίθεται αν κινδύνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια μέτρα bailout. Και θα πρέπει να κρίνει η σχετική αυτή Γενική Διεύθυνση αν οι δράσεις που θα εγκριθούν θα συνάδουν με τους κανόνες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή θα πρέπει να το κρίνει αυτό κάποια άλλη γενική διεύθυνση, δική σα γενική διεύθυνση. Πώς μπορούμε δηλαδή να αποφασίσουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποιος είναι υπεύθυνο για τις δύο αυτές σημαντικές αποφάσεις. Ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε εμείς να επαφιόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σημαντικές αυτές αποφάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Χρησιμοποίησα όντως κάποια αριθμητικά δεδομένα στην αρχική μου δήλωση. Τα αριθμητικά αυτά δεδομένα απορρέουν ουσιαστικά από τα δεδομένα τα οποία έχει δημοσιοποιήσει η Eurostat. Κάθε φορά, δύο φορές το χρόνο δεν κάνω λάθος, που η Eurostat κοινοποιεί τα δεδομένα για το χρέος και για το έλλειμμα, το κρατικό χρέος και το κρατικό έλλειμμα, υπάρχει πάντα και ένα παράρτημα, αυτό γίνεται από το 2008 και μετά, πάντα ένα παράρτημα λοιπόν, στα πλαίσια του οποίου βλέπουμε όλα αυτά τα αριθμητικά δεδομένα. και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να δούμε ξεκάθαρα πέρα από τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά δεδομένα ποια είναι τα έσοδα, ποιες είναι οι δαπάνες ενός, ενό, ενός κράτους, τι διακυβεύεται δηλαδή για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Και είναι πολύ σημαντικό να συνδυάζουμε τα δεδομένα αυτά με αυτά που έχουμε εμείς στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Όσον αφορά δηλαδή τα δημόσια αυτά κεφάλαια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να διασωθούν κάποιες τράπεζες, ε, Royal Bank of Scotland και άλλες. Έχουμε δηλαδή πολλές διαφορετικές πληροφορίες τις οποίες προσπαθούμε να συνδυάσουμε σε συγκεκριμένους ε, πίνακες προκειμένου να είναι πιο εύληπτες οι πληροφορίες αυτές και για τους ευρωβουλευτές αλλά και για οποιονδήποτε τελικά μεσολαβεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι εντυπωσιάζονται και ουσιαστικά πολλές φορές έχουν μια πάρα πολύ αρνητική άποψη για το τεράστιο αυτό ποσό το οποίο δόθηκε στο παρελθόν για να επιληθούν τα συστημικά προβλήματα των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν τα Χριστούγεννα λοιπόν υπόσχομαι ότι μέσω της Προέδρου σας ή άμεσα στα μέλη τη επιτροπή ΕΚΟΝ. Θα σα δώσω όλα αυτά τα αριθμητικά δεδομένα, όλου αυτού του πίνακες που θα σα βοηθήσουν να καταλάβετε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο θέσατε. Η οδηγία για την εκαθάριση των τραπεζών που βρίσκεται στα τελευταία στάδια τη ανάλυσή τη, είναι μια οδηγία που αφορά και τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θεσπίζει έναν κατάλογο bail-in για τις τράπεζες που βρίσκονται σε φάση εκαθάρισης, εξυγίανσης, δηλαδή τις μη βιώσιμες τράπεζες, αυτές οι οποίες πρέπει εις βάθος να αναδιαρθρωθούν, πρέπει να αλλάξουν επιχειρηματικό μοντέλο, πρέπει να αλλάξουν δομές και αρχιτεκτονική προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν στα πλαίσια της αγοράς. Η οδηγία στην υφιστάμενη κατάστασή της περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή έναν κατάλογο, αυτό το οποίο ονομάζουμε packing order στα αγγλικά, για τις τράπεζες δηλαδή εκείνες οι οποίες πρόκειται να συμμετάσχουν στο bail-in μιας τράπεζας που βρίσκεται σε φάση εξυγίανσης. Η λίστα λοιπόν είναι σύντομη γιατί βρισκόμαστε ακόμα σε μια φάση διαπραγμάτευσης της οδηγίας αυτής και η δική μας κατευθυντήρια γραμμή από πλευράς δηλαδή Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να έχουμε κατευθυντήρες γραμμές οι οποίες θα ισχύουν και για τις τράπεζες που βρίσκονται σε μια φάση ανακεφαλαιοποίησης, προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης. Δεν αναφέρομαι αυτή τη στιγμή σε μη βιώσιμες τράπεζες που βρίσκονται σε φάση εξυγίανσης, αλλά σε βιώσιμε τράπεζες οι οποίες βρίσκονται σε μια δύναμη αυτή τη στιγμή φάση και οι οποίες ενδεχομένως να χρειαστούν στο μέλλον ανακεφαλαιοποίηση. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν θα ήταν λογικό να χρησιμοποιήσουμε τις διατάξεις bail-in της οδηγίας. Ανταυτού έχουμε χρησιμοποιήσει το Ισπανικό Μνημόνιο του 2012 και προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα διαφορετικά στάδια ανακεφαλαιοποίησης και αναδιαργάνωσης των βιώσιμων τραπεζών, όπως για την SMS Real στις κάτω χώρες για την οποία πολύ σύντομα θα εγκριθεί ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης από τη στιγμή που θα έχουμε το απαραίτητο επίπεδο, επίπεδο κεφαλαίων. Η Ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει ένα bail-in για την βιώσιμη αυτή τράπεζα προτού αυξηθεί το κεφαλαίο της όπως αυτό το οποίο έγινε στο ισπανικό μοντέλο, στο ισπανικό παράδειγμα και το οποίο προβλέπεται και από τις κατευθυντήριες μας γραμμές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, ο κατάλογος αυτός αναγκαστικά πρέπει να είναι πιο σύντομος από τον κατάλογο εκείνο που προβλέπεται για τις μη βιώσιμες τράπεζες, οι οποίες θα μπουν σε μία φάση εξυγίανσης. Τώρα, τι θα γίνει για τη δεύτερη αυτή κατηγορία, τις τράπεζες αυτές οι οποίες πρέπει να εκαθαριστούν. Αυτό συζητούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμενη την οδηγία. Ποιος θα αποφασίσει τελικά αν η τράπεζα πρέπει να καθαριστεί, αν πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθεί. Και για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενδεχομένως να θέσουμε κατά μέρο τον κατάλογο των junior μετόχων και αυτών που διαθέτουν υβριδικά προϊόντα. Τον, τελευταίο, τον τελικό λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, αν πρέπει να καθορίσουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με ποιου τελικά θα μιλήσουμε. Με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα αναλάβει το λόγο του επιτηρητή στο νέο μηχανισμό που θα δημιουργηθεί. Ουσιαστικά θα μιλήσουμε με τη Φραγκφούρτη. Δεν απόκειται λοιπόν μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει αν υπάρχει κίνδυνος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αν οποιαδήποτε στιγμή υπάρξει μια αμφιβολία για την ερμηνεία του ενδεχομένου να παρουσιαστεί χρηματοπιστωτική αστάθεια, τότε θα ζητηθεί προφανώ και η γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν έχουμε, όπω είπατε, μια ιεραρχία και αποφασίσουμε κάποια στιγμή να μην ακολουθήσουμε την ιεραρχία αυτή, γιατί υπάρχει κίνδυνο χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θα έχει την πλήρη αρμοδιότητα αυτή, θα συζητήσει αποκλειστικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή θα εμπλακούν και άλλε γενικέ διευθύνσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω Γενική Διεύθυνση Μάρκτ. Κύριε Λάμπερτ, κοιτάξτε, πάντα συλλογικά 28 επίτροποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχουν στι συζητήσει αυτέ. Ο Επίτροπος Ανταγωνισμού είναι αυτός ο οποίος θα υποβάλει το αίτημα αυτό και στη συνέχεια με τη συμβολή των υπόλοιπων γενικών διευθύνσεων θα πρέπει να δούμε και τις τεχνικές πλευρές του φακέλου αυτού. Δεν μπορούμε εμείς όμως να λάβουμε μια πολιτική απόφαση. Έχουμε πολιτική απόφαση μόνο συλλογικά, όχι μεμονωμένα, συλλογικά ως Κολέγιο Επιτρόπων. Οι ερωτήσεις ε, αυτές για τις τράπεζες ε, τραβάνε. Ε, βεβαίως είναι πολύ επίκαιρο ζήτημα Προβλέπουμε όμως μία πιθανή αλλαγή θέματος γιατί θα περάσουμε στο ΕΛΚ και στον Ανδρέα Σουάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω και εγώ να αναφερθώ σε ένα ζήτημα της στιγμής που δεν είναι οι τράπεζες. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Επίτροπος στις αρχικέ του παρατηρήσεις. Τρία πράγματα θα ήθελα να πω. Ωραία. Τρία πράγματα θα ήθελα να πω. Πρώτα απ' όλα καλοδεχούμενα τα μνημόνια συνεννόησης με τις χώρες ε, BRIC και ελπίζω να μπορέσουμε να καλέψουμε όλες αυτές τις ε, χώρες έτσι ώστε η πολιτική του ανταγωνισμού να ε, εφαρμόζεται και να ελέγχεται παντού. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε γιατί χτες εδώ πέρα είχαμε μια συζήτηση για τον διαχωρισμό στην πρόταση που μας στείλατε μεταξύ ε, συλλογικών προσφυγών και της ε, πρότασης ε, για οδηγία και θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί τα έχετε διαχωρίσει, γιατί κάποιοι συνάδελφοι είναι υπέρ και δεν ξέρω αν εξακολουθεί να υποστηρίζετε το διαχωρισμό των δύο θεμάτων. Και τρίτον, το θέμα της Google. Ε, επιβεβαιώσατε στον κύριο Ραμόν Τρεμόζα πως δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια συνεννόηση, αλλά αν δούμε το πολύ πολύπλοκο αυτό ζήτημα με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους της αγοράς, ο ρωτάτε, ε, μήπως θα ήταν ευκολότερο να πάμε σε μια ρύθμιση των μηχανών αναζήτησης στην Ευρώπη αντί για ένα συμβιβασμό με τον κυρίαρχο παίκτη στην αγορά. Ίσως είναι κάπως ακαδημαϊκό το ζήτημα ή φιλοσοφικό, αλλά πρέπει να τεθεί, γιατί εμείς ως ευρωβουλευτές δεν ε, ξέρουμε τι συζητάνε οι υπηρεσίες σας με την Google και είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε τις λεπτομέρειες. Οπότε το ερώτημά μου είναι, θεωρείτε πως ε, πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση των μηχανών αναζήτησης στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κύριε Σφάμπ. Πρώτα όλα χαίρομαι για το ότι αναφέρεται το ζήτημα των BRICS, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στο Νέο Δελχή, στην Ινδία, όπου ήμουν στην τρίτη διάσκεψη των αρχών ανταγωνισμού των πέντε χωρών BRICS. Είναι σημαντικό να δούμε τι κάνουν αυτές οι ανερχόμενες οικονομίες και ανησυχούν ιδιαίτερα για την ε, ανάγκη ύπαρξης ισχυρών αρχών ανταγωνισμού και συγκλίνουν στα κριτήριά τους με τις ανεπτυγμένες χώρες και ειδικά πρέπει να σας πω πως οι περισσότερες από αυτές τις χώρες παρακολουθούν πάρα πολύ στενά το τι κάνουμε εδώ στις Βρυξέλλες, πιο στενά παρά το τι κάνουν ε, άλλες αρχές σε άλλα μέρη του κόσμου. Ακόμα και αν η συνεργασία ταξί ημών και άλλων συναδέλφων, ΙΠΑ, Αυστραλία, Κορέα κτλ. είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι λοιπόν ικανοποιημένος, αλλά ταυτόχρονα ανησυχώ γιατί υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών ε, με τις χώρες αυτές, ειδικά στον τομέα του ανταγωνισμού. Το πρώτο μνημόνιο συνεννόηση με τις χώρες αυτές νομίζω είχε υπογραφεί πριν από 10 χρόνια με μία από τις τρεις ε, αρμόδιες κινέζικες αρχές, το ε, Υπουργείο Εμπορίου. Τώρα έχουμε συμφωνία και με τις τρεις αυτές αρχές. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία λοιπόν με την ε, αρχή ανταγωνισμού στην Ρωσία μετά συζητήσαμε και τα της ε, Gazprom. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, ε, λέει ο κύριος Λάμπερτς. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ισχυρή. Κρίνουν 3.000 υποθέσεις το χρόνο. Ναι, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και ε, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Ανησυχούν ιδιαίτερα για τον κρατικό έλεγχο και είμαι ικανοποιημένο για το ότι το εξετάζουν αυτό. Βεβαίως, Έχουμε νέες σχέσεις με την αρμόδια αρχή της Κίνας, ε, της Βραζιλίας ε, και ο επόμενος στόχος μου ή δυνατόν πριν από τη λήξη της εντολής μας είναι να έχουμε ένα μνημόνιο συνεννόησης και με την νοτιοαφρικανική αρμόδια αρχή. Κατόπιν, εδώ πέρα πρέπει να ομολογήσω ε, στη, στην αίθουσα που δεν μας ακούει κανείς. <laughs> Η πρόεδρος λέει μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Πώς ε, απογοητεύομαι από τον ε, κίνδυνο καθυστέρησης που υπάρχει, από το πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα της ε, οδηγίας περί ιδιωτικής δράσης. Θυμάμαι εδώ πέρα όταν είχα την πρώτη φορά στην ακροασή μου και είπα πώς ε, θα προσπαθήσω να προωθήσω νομοθεσία ιδιωτικής επιβολής του, ε, της νομοθεσίας. Και είχαμε πράγματι καταλήξει στο διαχωρισμό της ε, συλλογικής ε, πρόσφυγης και τη, από την ιδιωτική επιβολή και τελικά το δέχτηκα για να έχουμε μια θετική απόφαση του Κοινοβουλίου εντός της θητείας αυτής υπέβαλα μία πρόταση, δηλαδή το Σώμα των Επιτρόπων, με κάποια συμπληρωματικά στοιχεία μη νομικής φύσης για τις ε, συλλογικές προσφυγές, για να προωθηθεί η συζήτηση, για να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν εθνική νομοθεσία. Και όταν θεωρούσα πως ε, οι πιο δύσκολες συζητήσεις θα ήταν στο Συμβούλιο, διαπιστώνω πως το Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα κατά 99% θα πάω στο γιους τους λήψους και θα υπάρχει συμφωνία για τη γενική προσέγγιση σε πρώτη ανάγνωση, εδώ πέρα έχω σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα προλάβει το Κοινοβούλιο. Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους εσάς και ιδιαίτερα τον κύριο Σβάμπ, τον εισηγητή, να με βοηθήσετε να έχουμε μια καλή συζήτηση εις βάθος για να έχουμε μια ευτυχή κατάληξη της υπόθεσης πριν λήξει η θητεία σας. Όχι η δική μου θητεία, θα έχω κάποιους μήνες ακόμα, αλλά πριν λήξει η δική σας θητεία. Όσον αφορά την Google, ε, κάτι ακόμα. Για να... Απαντώντας τον κύριο Φάλμπα είπα πως θεωρώ μαζί με τον Μισελ Μπαρνιέ πως το θέμα των ΜΥΦΣ κάποια στιγμή χρειάζεται κάποια ρυθμισή. Είμαι σοσιαλδημοκράτης δεν ε, υπάρχει νομίζω υποψία. Μα έχουμε δει τέτοιους σοσιαλδημοκράτες που κάνουν αυτά τα οποία λέτε. Εγώ δεν είμαι ούτε το ένα ούτε το άλλο όμως, λέει ο κύριος Επίτροπος. Είμαι κάπου στο κέντρο της σοσιαλδημοκρατίας όσον αφορά την αξία της ρύθμισης δηλαδή. Αλλά, ειλικρινά, δεν βλέπω ανάλυση να δικαιολογεί ρύθμιση των μηχανών αναζήτησης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση, πάρα πολύ εκφέρουν άποψη, άλλοι αιτιολογημένοι, άλλοι όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας μπορεί να πει ε, ότι θεωρεί σωστό. Είναι η έρευνα περίπλοκη και δεν μπορώ να προβλέψω πώς από αυτή την περιπλοκότητα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κανονισμό. Όχι ακόμα. Ίσως στην επόμενη θητεία. Σας ευχαριστώ. Αλλάζουμε τώρα την ε, σειρά. Αντώνιο Κένσια, νομίζω παρέφθηρα δολοφόνησα το όνομά σας, αλλά μπορώ να το κάνω γιατί είμαι πρόεδρος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο. Θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στις κρατικές ενισχύσεις, αν θέλετε. Πιστεύω ότι όσο έχει ε, η κατάσταση αυτή τη στιγμή, ιδίως μετά την απόφαση για το αεροδρόμιο της Λιψίας, Θεωρώ ότι υπάρχει μια κάποια σύγχυση αυτή τη στιγμή για το όλο πλαίσιο το οποίο διέπει τις κρατικές ενισχύσεις. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο. Εν γέννη, αν κρατική ενίσχυση τελικά σημαίνει οποιαδήποτε συμμετοχή σε μια οικονομική δραστηριότητα, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα θέσουμε πραγματικά σε κρίση το όλο σύστημα σύμπραξης και συνεργασίας ιδιωτικού δημοσίου τομέα, γιατί ξέρετε ότι ο ιδιωτικό τομέα συμμετέχει σε μια οικονομική δραστηριότητα και προφανώς από την οικονομική αυτή δραστηριότητα ο ιδιωτικό τομέα θέλει να κερδίσει και κάποια χρήματα. Διαφορετικά δεν υπάρχει κανένα κίνητρο συμμετοχή του. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν γενικό είναι το ακόλουθο. Πραγματικά θέλουμε με το σύστημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουμε εν κινδύνο το μόνο σύστημα, δηλαδή τη σύμπραξη ιδιωτικού, ιδιωτικού δημοσίου τομέα, το μόνο σύστημα το οποίο λειτουργεί καλά αυτή τη στιγμή για τι επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, όσον αφορά γενικότερα την κατασκευή υποδομών, τα έργα υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρομαι ακόμα και στις πολιτιστικές υποδομές, δηλαδή στην κατασκευή μουσείων και το διανύουμε μία περίοδο όπου τελικά πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Πέρα από τις αποφάσεις για τα ευρυζωνικά δίκτυα ή για τα αεροδρόμια ή ενδεχομένως και για τους λιμένες αργότερα, για την υδρολεκτρική ενέργεια για παράδειγμα ή για τον μουσιακό τομέα. Για όλους αυτούς λοιπόν τους τομείς όπου έχουμε πολύ σημαντικές υποδομές θα έχετε ξεχωριστό καονισμό για κάθε τομέα και για κάθε υποδομή ή θα προχωρήσετε σε μια γενική ρύθμιση, σε ένα γενικό κανονισμό και θα διευκρινίσετε κάπως καλύτερα τι εννοείται όταν χρησιμοποιείτε τον όρο κρατική ενίσχυση. Ξέρετε ότι ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες αυτή τη στιγμή συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς και πολύ φοβάμαι ότι ε, ενδεχομένως να θέσετε εν κινδύνο με τους κανονισμούς σας διαγωνισμούς που έχουν ήδη ξεκινήσει και προτάσεις συμμετοχής που ήδη έχουν γίνει, αιτήσει συμμετοχής που έχουν ήδη γίνει από την ιδιωτικό τομέα. Φοβάμαι αυτή τη στιγμή ότι προχωράμε σε ένα κλίμα πάρα πολύ μεγάλης σύγχυσης, ακόμα και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Βλέπω ότι τα πάντα αυτή τη στιγμή συζητώνται από την αρχή. Και αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι κατά περίπτωση μόνο λαμβάνονται κάποιες μονομένες αποφάσεις χωρίς να μπορούμε πλέον ως κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζουμε τελικά αν ισχύει ένας γενικός κανόνας ενιαίος για όλους, όσον αφορά δηλαδή το τι είναι κρατική ενισχύση και το τι δεν είναι. Θα μπορούσατε λοιπόν κύριε Επίτροπε να μην ενημερώσετε λίγο επ' αυτού, να με διαφωτίσετε λίγο περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα είναι πολύπλοκο εγχείρημα το να ελέγχει κανεί τι κρατικέ ενισχύσει και κάθε φορά που υπάρχει μια απόφαση από το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πρέπει εμεί να αναλύουμε την απόφαση αυτή και να δούμε τελικά αν η νομολογία του δικαστηρίου τελικά συνάδει με τις δικές μας κατευθυντήριες γραμμέ, με το δρόμο τον οποίο ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας δούμε πως έχουν βελτιώσει όμως οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γενικότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ήδη από τη συνθήκη της Ρώμης και μετά έχουν γίνει πάρα πολλά θετικά πράγματα. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το μέσο αυτό, γιατί μέσω αφού του μέσου καταφέρνουμε τελικά και βελτιώνουμε τα κριτήρια τα οποία εμείς χρησιμοποιούμε για τις κρατικές ενισχύσεις. Ξέρετε ότι μέσω της νομολογίας του δικαστηρίου μπορούμε εμείς να αποφασίζουμε στη συνέχεια για συγκεκριμένους κανόνες, συγκεκριμένες άδειες, συγκεκριμένους περιορισμούς. Αναφερθήκατε τώρα στην δικαστική απόφαση όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για το αεροδρόμιο της Λειψίας. Προφανώς πρέπει εμείς να λάβουμε υπόψη μας στη σχετική νομολογία βασίζεται σε συγκεκριμένη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα όμως από την απόφαση αυτή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ε, υπόλοιπες διαφορετικές περιπτώσεις, τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, να δούμε τις καταγγελίες που γίνονται από τα ίδια τα κράτη-μέλη και να δούμε αν εξ ε, υπάρχει παραβίαση των υφιστάμενων κανόνων. Τώρα, αν έχουμε μια εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα, όπως είπατε, προφανώς έχουμε τότε εμπλεκόμενους από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που συμμετέχουν και επενδύουν σε ένα επίπεδο. Αν λοιπόν συμμετέχουν και συνεργάζονται με αυτόν τον τρόπο και επενδύουν ισότιμα, σε ισότιμε συνθήκε, τότε δεν υφίσταται καν η έννοια τη κρατική ενίσχυση. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί έχουμε ισότιμου όρου ανταγωνισμού. Αν όμω έχετε μία σύμπραξη, μία εταιρική σχέση δημοσίου, ιδιωτικού τομέα, όπου όλη την ευθύνη και όλο το βάρο ευθύνη φέρει ο δημόσιο τομέα, ε, ενώ ο ιδιωτικό τομέα δεν φέρει κάποια ευθύνη, ή το αντίστροφο, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε στη δεύτερη αυτή περίπτωση για κρατική ενίσχυση εφόσον ο ιδιωτικό τομέα που αναλαμβάνει όλη την ευθύνη. Σα το λέω αυτό για να σα πω ότι πρέπει στι περιπτώσει αυτέ να εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και ξέρετε ότι και τα κριτήρια μπορούν να είναι διαφορετικά. Όταν εξετάζουμε για παράδειγμα τις δημόσιες επενδύσεις για τις υποδομές, τα πράγματα τώρα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια, όταν δεν είχαμε όλη αυτή τη σορευμένη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε να μεταφράσουμε τώρα τα κριτήρια της συνθήκης στην πράξη και πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς μπορούν οι αποφάσεις αυτές να γίνουν κατανοητές για αυτούς οι οποίοι σε καθημερινή βάση και χωρίς να έχουν όλη τη νομική εμπειρογνωμοσύνη πρέπει να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου και τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα πακέτο απλούστευσης όσον αφορά τους κανόνες αυτούς και θέλουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή έννοια και ένα κοινό ορισμό όσον αφορά την κρατική ενίσχυση. Δεν μπορούμε εμείς όμως να δημιουργήσουμε από το μηδέν τον ορισμό αυτό θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτό το οποίο ήδη υφίσταται και να καταφέρουμε τελικά να αποσαφηνίσουμε και να απλουστεύσουμε το τι είναι κρατική ενίσχυση βασιζόμενη στα όσα μας έχει ήδη πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βασιζόμενο δηλαδή στον ορισμό που το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δώσει μέχρι στιγμής και όλα αυτά τα χρόνια στην έννοια τη κρατική ενίσχυση. Όταν θα έχουμε ήδη προετοιμάσει μια πρόταση και ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προφανώ θα συνεργαστούμε μαζί σα για να βελτιώσουμε το κείμενο αυτό. Τώρα, υπάρχουν ορισμένε υποδομέ από την άλλη, που κατά την άποψή μα αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση από ό,τι είναι για παράδειγμα τα αεροδρόμια στα οποία αναφερθήκατε, οι πολιτιστικές υποδομές, οι υποδομές του πολιτιστικού τομέα που δεν παρέχουν αναγκαστικά μια υπηρεσία στην αγορά, αλλά παρέχουν μια υπηρεσία την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε πιο κρατική, πιο δημόσια, μια πιο κεντρική υπηρεσία αν θέλετε. θα έχουμε έναν κανονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προβλέπει συγκεκριμένε εξαιρέσει για τις υποδομές αυτές και ο οποίος θα διαφέρει τελικά από τον κανονισμό του 2005 όσον αφορά τις εξαιρέσει για τις κρατικές ενισχύσεις. Τώρα, Όσον αφορά τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, ξέρετε ότι εγκρίναμε ένα κείμενο στα τέλη του 2012 και ελπίζουμε ότι στα μέσα του 2014 θα έχουμε μια οδηγία για την έρευνα και την καινοτομία και μια οδηγία για την ενέργεια και το περιβάλλον. Το ζήτημα λοιπόν των υποδομών για την έρευνα και την κεντομία θα μας απασχολήσει, καθώς επίσης και οι υποδομές για το περιβάλλον και την ενέργεια. Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι την υφιστάμενη νομολογία του δικαστηρίου, προκειμένου να προσδώσουμε στα κείμενα αυτά την υψηλότερη δυνατή νομική βεβαιότητα. Κάθε φορά που πρέπει δηλαδή να αποφασίζουμε τι είναι κρατική ενίσχυση και τι όχι. Τώρα, αν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο μία υπόθεση πηγαίνει στο δικαστήριο και πρέπει να εκδικαστεί ζήτημα ανταγωνισμού και κρατικής ενίσχυσης, τότε αναγκαστικά εργαζόμαστε αναπερίπτωση. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια ελάχιστα πρότυπα τα οποία ήδη ισχύουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα οποία μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση και έχουμε έπειτα τον καονισμό με τις γενικές εξαιρέσεις, ο οποίος ε, μας βοηθά να αποφανθούμε για το ότι ναι, όντως κάτι είναι κρατική ενίσχυση, αλλά δεν υπήρξε εκ των προτέρων κοινοποίηση. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, καλούνται οι εμπλεκόμενοι να ακολουθήσουν τις κανόνες και θα έχουν κάποιες επιπτώσεις αν δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες αυτούς. Και έπειτα υπάρχει και ένα όριο πάνω από το οποίο καλούμεθα να εξατάσουμε κάποιες περιπτώσεις εντελώς ξεχωριστά, τις περιπτώσεις εκείνες όπου φοβόμαστε τελικά ότι υπήρχε κρατική ενίσχυση ενώ την επιτρεπότανε. Βασιζόμαστε λοιπόν στην ομολογία του δικαστηρίου όπως καταλάβατε, αλλά πάντα θα υπάρχει μια σαφής γκρίζα ζώνη την οποία θα καλούμε θα να αναλύσουμε προτού πάρουμε μια τελεσίδικη απόφαση. Ξέρετε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει να γίνονται προσφυγές κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να αποσαφινιστούν κάποιες περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων. Eh. Ευχαριστώ που ήρθατε Επίτροπε. Θα ήθελα να μου κάνετε μία διευκρίνηση σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση. Θα ήθελα Λοιπόν, ω προ την ε, Τραπεζική Ένωση, να ε, ε, συμπληρώσετε κάποια στοιχεία στην προηγούμενη παρέμβασή σα, όπου περιγράψατε τι βασικέ αρμοδιότητε κυρίω για τη μεταβατική περίοδο, μέχρι ότου τεθεί σε ισχύ και αρχίσει να λειτουργεί ο ενιαίο υποπτικό μηχανισμό. Λοιπόν, αν ο βασικό στόχο είναι η σταθερότητα, η ολοκλήρωση τη αγορά και η προστασία των καταναλωτών, θα πρέπει να κινηθούμε ταχύτατα. Αυτό θα είναι δυνατόν ακόμη ε, και δεδομένης της τωρινής συγκυρίας. Στη συνέχεια, ως προς την ολοκλήρωση των αγορών. Ε, οι λύσεις που θα υιοθετηθούν θα είναι εξισορροπημένες ε, όπως στην περίπτωση του ανταγωνισμού. Γιατί είδαμε τι συνέβη στην Ισπανία και αναρωτιόμαστε αν θα προβλεφθούν επαρκείς διατάξεις. Κατόπιν, για την ανακεφαλαιοποίηση, αν πραγματοποιηθεί με δημόσια κεφάλαια, τι ακριβώς ε, θα συμβεί ε, με τις αποκρατικοποίησεις ε, θα ανακτηθεί ένα μέρος από αυτά τα δημόσια κεφάλαια. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ερμηνεύσει τις προθέσεις του Κοινοβουλίου είναι αναμφισβήτητη η βούληση του Κοινοβουλίου να αντεπεξέλθει στις τωρινέ προκλήσεις και χρειαζόμαστε μια ισορροπία ανάμεσα ε, στα προγράμματα και τους στόχους ε, που έχουμε θέσει. Τα προγράμματα λοιπόν επί σε, σε ποιο βαθμό ε, χρειάζονται για, να, ε, για τη δίωξη των καρτέλ, των συμπράξεων. Έχετε στοιχεία να μας δώσετε για αυτά τα προγράμματα επί οίκιας, επικού μεταχείρισης στα πλαίσια της επιβολής κυρώσεων των καρτέλ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας δω, ε, διευκρινίσω ότι οι κατευθυντήριες γραμμές ε, για την ε, ασφάλεια κατά τη μεταβατική περίοδο ο στόχος είναι να διευκολύνουν τη μεταβατική περίοδο αλλά εξαρτάται Βεβαίω και πόσο θα κρατήσει η μεταβατική περίοδο. Θα πρέπει να δούμε όλα τα επιμέρους στοιχεία της ε, ασφάλειας ε, στον τραπεζικό τομέα. Αυτό που δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ε, Τραπεζικής Ένωσης είναι να έχει αποκλειστική αρμοδιότητα ε, να μην έχει μάλλον αποκλειστική αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον έλεγχο των κρατικών επιδοτήσεων. Αυτό αναγράφεται στι συνθήκε και ουδή ε, το αμφισβητεί. Ουδή αμφισβητεί επίση ε, τι υπόλοιπε αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Γιατί σε περιπτώσει, ε, τι κατεπίγουσε περιπτώσει και δυστυχώ βιώσαμε τέτοιε περιπτώσει από την απαρχή τη κρίση μέχρι σήμερα, από νυχθημερών είδαμε ότι ε, κάποιες τράπεζες ε, βρέθηκαν σε πλήρη αδυναμία να αντιμετωπίσουν την πίεση των αγορών. Ε, δεν είχαν καθόλου κεφάλαια στη διάθεσή τους και από τη μία μέρα στην άλλη λοιπόν χρειάστηκαν μία πάρα πολύ σημαντική ένεση κρατικών κονδυλίων. Τι θα γίνει λοιπόν ε, χρειάζεται, όπως και ε, από τότε που άρχισε η κρίση, να λαμβάνει εξαιρετικά περίπλοκες αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρα πολύ γρήγορα και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει ε, σωστές αποφάσεις με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε δεν να μην επαναληφθούν αυτές οι περιπτώσεις ή τουλάχιστον να είναι πιο περιορισμένης εμβέλειας ε, σε σχέση με αυτά που ζήσαμε όλοι το 2008. Σε κάθε περίπτωση ε, η επικοινωνία ανάμεσα στον ενιαίο επόπτη και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή ας το πω διαφορετικά ε, η επικοινωνία ανάμεσα στην αρχή αρμόδια για τον έλεγχο των κρατικών επιδοτήσεων και ε, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που εν μέρη θα έχει τις αρμοδιότητες του ενιαίου απόπτη έχει ιδιαίτερη σημασία. Ε, ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα γιατί δεν, ήδη το, έχουμε, έχουμε αναλάβει τέτοιο ρόλο το ζήτημα που τίθεται είναι ότι κάποια κράτη-μέλη και ελπίζουν να μην επαναληφθούν αυτές οι περιπτώσεις ε, και ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες ε, ε, εκεί που πρέπει στην Ευρωζώνη. Κάποια κράτη-μέλη λοιπόν επιτυχώς κατάφεραν να περάσουν το μήνυμα ότι ένα ε, μικρό πρόβλημα της οικονομίας τους ε, έχει ε, συστημική σημασία. Και τελικά δεν εφαρμόζουμε τους κανόνες, αλλά εφαρμόζουμε τις εξαιρέσεις. Γι' αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων περιπτώσεων προσπαθούμε το νέο σύστημα να εδράζεται επί κρατεότερων πυλώνων αν θέλετε και ε, το προηγούμενο σύστημα δεν μπόρεσε να ε, ρυθμίσει την κατάσταση λόγω της ε, μεγάλης συγκέντρωσης προβλημάτων στην Ευρωζώνη. Ξαναλέω ότι ελπίζω να μην επαναληφθούν αυτά στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, αν διαπιστώνουμε ότι απειλείται η μακροοικονομική σταθερότητα από τέτοιες απειλές, Ε, θα ε, εστιάσουμε τις συζητήσεις μας γύρω από τον μηχανισμό ε, ταχείας αντίδρασης ε, αλλά ε, ξαναλέω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Δεν μπορεί οι πολίτες να ε, βλέπουν ότι αυτό πλέον συνιστά τρέχουσα πρακτική και αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζητάμε από τους πολίτες να αδειάζουν τις τσέπες τους για να βρουν τα τελευταία σέντια να στηρίξουν και πάλι τις τράπεζες αυτοί που πρέπει να επέμβουν είναι αυτοί που ε, είναι ε, ε, μέσα στο σύστημα οι πιστωτές, οι πελάτες των τραπεζών, οι μέτοχοι των τραπεζών. Με ιδιαίτερα πειθαρχημένο και διαφανή τρόπο θα πρέπει να οργανώσουμε λοιπόν τις εργασίες μας, θα πρέπει να ε, επικοινωνούμε με εσάς αλλά και με τους πολίτες ε, εν μέρη αποκρατικοποίησης και εν μέρη ενέσεις και άλλων δημοσίων κεφαλαίων ε, μπορεί να συμβούν και στο μέλλον. Ε, υπήρχαν περιπτώσεις όπου ε, υπήρχε δημόσια συμμετοχή σε μια τράπεζα ε, η οποία όμως ε, απεσύρθη και ανακεφαλοποιήθηκε η τράπεζα με χρήματα των φορολογουμένων. Αυτή η πυραμίδα όμως που είχε δημιουργηθεί έχει καταρρεύσει σε μεγάλο βαθμό και τελικά εδόθηκε μόνο το 1 τρίτο των προεξεγγελθήσεων εγγυήσεων και τελικά συνειδητοποιούμε πως ε, έχουμε πληρώσει ήδη ε, για τις επιπτώσεις ε, του συστήματος που είχαμε επιλέξει στο παρελθόν και τελικά Υπήρξε μία περίοδος από το 2010 μέχρι το 2012 όπου μειώθηκαν οι εγγύησεις κατά δύο τρίτα. Εγώ πιστεύω ότι τελικά γίνονται οι απαιτούμενες οικονομικές προσαρμογές αλλά ε, ε, ακόμη έχουμε πάρα πολλές απειλές ε, για τους φορολογούμενους. Δηλαδή τι σημαίνει μια κρατική εγγύηση. Αυτή η κρατική εγγύηση αποζημιώνεται με κάποιο τρόπο και το εισόδημα μπαίνει στον προϋπολογισμό του κράτους. Ε, ε, στη συνέχεια η εγγύηση η οποία χρησιμοποιείται στην τράπεζα μπαίνει στα περιουσιακά στοιχεία της ε, τράπεζας και άρα προκύπτουν και μερίσματα από αυτή. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και έσοδα από αυτό, 125 συγκεκριμένα εισόδημα για τα τα κράτη-μέλη. Ε, όμως, δεδομένου του κινδύνου που διέτρεξαν τα κράτη-μέλη και οι πολίτες, ε, είναι αμεληταίο το πόσο ε, για τα προγράμματα επίοικους μεταχείρισης. Σας είπα ήδη κάποια πράγματα και νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σε μια πιο στοχευμένη συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Κλείνω σχεδόν τέσσερα χρόνια στη θέση του Επιτρόπου Αρμοδίου για τον Ανταγωνισμό και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε λειτουργήσουν ε, εύρυθμα αυτά τα προγράμματα επί οίκες. Ε, ουδάλλως ε, η καταπολέμηση, ο αγώνας μας κατά των συμπράξεων των καρτέλ θα υπονομευθεί. Δεν μπορούμε να πούμε παραδείγματος χάρη ότι μία επιχείρηση η οποία έχει μετάσχει στο παρελθόν σε ένα καρτέλ αυτή η μεταχείριση ε, ε, θα απαλλαγεί από την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης ε, στο μέλλον. Ξαναλέω ότι είναι απαραίτητο το πρόγραμμα για την καταπολέμηση των καρτέλ. Ευχαριστούμε. Μπέρτολ τώρα από το ΕΛΚΑ. Okay. errori di Άκουσα κύριε Επίτροπε, την παρουσίαση που κάνατε και θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά είναι λίγο ωριακό θα έλεγα. Βρίσκεται στα όρια ανάμεσα στη δική σας αρμοδιότητα και στην αρμοδιότητα κύριου Μπαρνιέ. Αναφέρομαι στις εκχωρήσεις. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλα τα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουν να απελευθερωθούν οι απαραίτητοι πόροι για να έχουμε επενδύσεις για μεγάλα δημόσια έργα. Και ξέρουμε ότι πολλές από τις επενδύσεις αυτές τελικά χρηματοδοτούνται μέσω των εταιριών εκείνων των ιδιωτικών που συμμετέχουν σε εκχωρήσεις και οι οποίες τελικά χρηματοδοτούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δημόσια έργα μέσω της συμμετοχής τους σε δημόσιους διαγωνισμούς. Αλλά όταν οι ιδιωτικές αυτές εταιρείες πολλές φορές βρίσκονται πολύ κοντά στην λήξη της χρονικής αυτής περίοδου της εκόρησής τους, δεν μπορούν να δώσουν τις απαραίτητες τραπεζικές εγγυήσεις με αποτέλεσμα να σταματά το έργο μετά. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε τα απαραίτητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επιτρέπουν ε, την παράταση τη χρονική της εκχώρησης έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί σωστά το δημόσιο αυτό έργο και να δοθούν οι απαραίτητες τραπεζικές εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση του έργου αυτού. Κατά αυτόν τον τρόπο, μέσω της παράτασης αυτής της χρονικής θα απελευθερωθούν περισσότεροι πόροι οι οποίοι είναι ουσιαστικά διαθέσιμοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τελικά ανταποκρίνονται στις επενδύσεις που μπορούν άμεσα να γίνουν γίνουν επενδύσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από μια επίσημη διαδικασία διαγωνισμού και οι οποίες όμως δεν μπορούν, οι πόροι αυτοί δεν μπορούν να δοθούν ακριβώς επειδή τελειώνει η περίοδος εκχώρησης και δεν μπορούν να δοθούν οι απαραίτητες τραπεζικές εγγύσεις. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όπως το είπατε, είναι ο κύριος Μπαρνιέ που είναι πιο αρμόδιος για τα ζητήματα αυτά. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς εν γέννη. Είναι ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς αυτός ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει πρόταση νομοθεσίας για τον τομέα αυτό. Η δικιά του Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για το ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε. Τώρα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις εκχωρήσεις αυτές, όταν δηλαδή έχουν εγκριθεί στα πλαίσια ενός δημόσιου διαγωνισμού, το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να εμφανιστούν φαινόμενα κατάχρησης, ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες έμεσες κρυφές κρατικές ενισχύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές θα έπρεπε εγώ τότε να δω τι ακριβώς συμβαίνει, να αναλύσω την κατάσταση και να λάβω κάποια μέτρα. Δεν ξέρω αν σε όλες τις περιπτώσεις θα καταλήξουμε σε έρευνα, πάντως να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχουμε μία περίπτωση όπου σε μία χώρα πρόκειται να παραταθεί η περίοδος εκχώρησης, χωρίς όμως να έχει τελικά γίνει επίσημος διαγωνισμός χωρίς να έχουν ε, μπορέσει και άλλες ιδιωτικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην όλη αυτή διαδικασία. Αν λοιπόν στην περίπτωση αυτή λάβετε εσείς μια απόφαση για χρονική παράταση, η οποία ευνοεί μία και μοναδική μόνο εταιρεία, τότε καταλαβαίνετε ότι ε, στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένας μόνο φορέας, ο οποίος θα ευνοηθεί χρηματικά και τότε μιλάμε για μία κρυφή έμεση περίπτωση κρατικής ενίσχυσης ή ενδεχομένως μέσω του συστήματος αυτού να προβλέπεται μια κάποια αποζημίωση για μια οικονομική υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος. Και στην περίπτωση αυτή πάλι θα πρέπει να δούμε ποια ήταν η αρχική διαδικασία διαγωνισμού, αν όντως δηλαδή τα πάντα έγιναν με απόλυτη διαφάνεια ή αν υπήρξε μια κάποια χειραγώγηση. Πάντως, από νομοθετικής πλευράς το παραλαμβάνω ότι δεν είναι η δική μου γενική διεύθυνση η οποία μπορεί να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Πρέπει πρώτα να γίνει μια νομοθετική πρόταση από τη Γενική Διεύθυνση του κ. Μπαρνιέ και εμείς στη συνέχεια θα δούμε αν οι κανόνες στηρούνται. Κυρία Στάλερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, άλλοι μίλησαν για τα επίκαιρα. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι η κυβέρνηση της Σκωτίας σήμερα δημοσίευσε μια λευκή βίβλο για την ανεξαρτησία της Σκοτίας και λέει κάποια πράγματα για, την, για τις σχέσεις της ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Εθνικό Σκοτσέζικο Κόμμα λέει πως θα χρησιμοποιήσει το άρθρο 40, ότι δεν θα είναι δηλαδή μια τυπική διαδικασία Ενταξύ θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις εξαιρέσεις που υπάρχουν ήδη για το ευρώ, τη ζώνη Σέγγεν και να διατηρήσουν και ένα κομμάτι της Βρετανικής επιστροφής. Θεωρούν πως η Σκοτία μέχρι τις 24 Μαρτίου 2006 θα είναι το 21ο κράτος μέλος. 18 μήνες δηλαδή μετά το δημοψήφισμα. Θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας. Μπορεί μια νέα χώρα να ενταχθεί στην Ένωση χωρίς να περάσει από τη διαδικασία ένταξης και να δεσμευτεί να μπει στο ευρώ και έχει λάβει ποτέ ένταξη χώρα σε 18 μήνες. Έχει. Σας ευχαριστώ. Προσπαθώ να βρω κάποια σχέση μεταξύ της ερώτησής σας και των αρμοδιοτήτων μου. Δεν μπόρεσα βεβαίως. Όχι, όχι, περιμένετε. Περιμένετε κύριε Λάμπερτς. Εν πάση περιπτώσει, είμαι μέλος της Επιτροπής, πολιτικός Τι θα γινόταν εάν το ερώτημα αυτό απευθυνόταν προς τον έναν υπεύθυνο να απαντήσει. Θα σας πω τι θα ήθελα εγώ να απαντήσω υπεύθυνο. Θα έλεγα πως η θέση μου πριν να είναι πολύ αργά είναι να ενθαρρύνω τους Σκοτσέζους να ψηφίσουν κατά της ανεξαρτησίας και δεύτερον εάν δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι υπέρ της ανεξαρτησίας. Δυστυχώς θα ανακαλύψουν οι υπέρμαχοι του ναι πως α, το επόμενο λεπτό θα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω πως είναι σαφές. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε και νομίζω εδώ πέρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Ναι κύριε Λάμπερτς. Νομίζετε πως υπάρχει ζήτημα ανταγωνισμού μεταξύ Σκοτίας, Καταλωνίας, Φλάνδρας, Παδανίας για να κλείσουν, ξέρω εγώ, ημερομηνία δημοψηφίσματος. Η απάντηση του Επιτρόπου είναι πως βεβαίως εσείς ως Βέλγος δεν μιλάτε για τις κοινότητες αλλά μόνο για τις περιφέρειες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα διακόψουμε για λίγο και μετά θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. So, seguimos con el orden del día, que es el punto 13 de la agenda. Περάσουμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Εξέταση του σχεδίου για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια της κυρίας Κράτσα που είναι παρούσα. Παρακαλώ, δίχως περαιτέρω καθυστέρηση, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ήθελα καταρχάς να πω ότι η προσέγγιση μου προς την πρόταση της Επιτροπής είναι θετική. Είναι η δεύτερη φορά που συζητούμε το θέμα και έχει γίνει και μια δημόσια ακρόαση η οποία ήταν πολύ ωφέλιμη για την ε, υπόθεση που επιρετούμε. Η προσέγγιση μου είναι θετική διότι είμαστε πια, η πρόταση αυτή έχει να κάνει με τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης της οικονομίας και έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει ένα είδος από αυτές τις μορφές. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι συζητούμε για μακροπρόθεσμα, ε, μακροπρόθεσμη δυνατό, ένα σχήμα για μακροπρόθεσμες δυνατότητες ε, επενδύσεων, κάτι στο οποίο πάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και έρχεται η πρόταση της Επιτροπής να δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο θα έχει ένα ευρωπαϊκό χαρακτήρα με, τον, με την έννοια ότι θα δίνει μια ασφάλεια προς τους εγχώρους και ξένους επενδυτές ότι είναι κάτι συγκεκριμένο, σαφές, αναγνωρίσιμο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι θα ενθαρρύνει την, ε, όχι μόνο τη δραστηριοποίηση ευρωπαϊκών κεφαλαίων αλλά και ξένων εκτός Ευρώπης επενδυτών και θα δώσει αυτή την ε, ζωντάνια στις διασυνοριακές ε, δραστηριότητες. Επιπλέον, είναι κάτι το οποίο ε, στοχεύουμε να δώσει τη δυνατότητα σε μικροεπενδυτές να επενδύσουν. Σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχουν χρήματα, παρόλη την οικονομική κρίση και τις συνέπειές της στην κοινωνία, υπάρχουν χρήματα εκτός τραπεζών που περιμένουν να δούνε πού μπορούν να πάνε. Ε, οι, οι, οι συμπολίτες μας ανησυχούν για την εξέλιξη των συνταξιδοτικών του συστημάτων, θα θέλαν να έχουν κάτι σαφές και ασφαλές για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, είναι μια, μια ε, έξοδος σε αυτές τις ανάγκες το, το νέο ταμείο το οποίο έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει. Οι τροπολογίες οι οποίες κατέθεσα έχουν να κάνουν καταρχάς με την ενθάρρυνση του να, των, ο, επενδύσεων ε, στις εισηγμένες ε, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο από όσο ήδη δίνει το σχήμα το που προτείνεται. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι στο κομμάτι του 75% επιλέξιμων δαπανών επενδύσεων από το, χαρτοφυλάκιο. Αφενός γιατί και οι μικρομεσαίες εισηγμένες έχουν και αυτές ανάγκη ανάγκη χρηματοδότησης, αλλά και αφετέρου ο, ε, είναι, ε, δίνουν την ασφάλεια και τη διαφάνεια του χρηματιστηρίου. Πιστεύω ότι για να γίνει ελκυστικό το σχήμα αυτό, διότι για να πετύχει το στόχο του πρέπει να είναι ελκυστικό στην αγορά. Για να είναι ελκυστικό, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τον κύκλο ζωής των ταμείων αυτών, ο οποίος θα έχει βέβαια μια συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν μπορεί να είναι κάτι ανοιχτό παόριστον, αλλά μπορεί να έχει τη δυνατότητα να το επεκτείνει ή να το λήξει νωρίτερα ο διαχειριστής όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες. Παραδείγματο χάρη ένα project χρειάζεται περισσότερο χρόνο ή ένα τέτοιο σχήμα είναι γενικότερα επιτυχημένο και κερδοφόρο. Κάτι άλλο που με απασχόλησε ιδιαίτερα είναι οι δυνατότητες ε, των μικροεπενδυτών που μπορούν να έχουν κάποια ευελιξία δηλαδή, διότι είναι γεγονός ότι το πολύ μακροπρόθεσμο σχήμα δεν είναι γενικά ευνοϊκό για αυτούς. Έτσι πιστεύω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα αναφέρονται ε, συγκεκριμένα στο καταστατικό του νέου σχήματος, ε, μπορούν να έχουν τη δυνατότητα εξαγοράς του μεριδίου τους, μικρού μεριδίου και με προϋποθέσεις όπως είπα, ή μπορούμε να δούμε και θα ήθελα και την ε, γνώμη των συναδέλφων για τη δυνατότητα μεταβίβασης του μεριδίου, αν όχι εξαγοράς, μεταβίβασης του μεριδίου, εν πάση περιπτώσει μια μορφή ε, ευελιξίας για τους μικροεπενδυτές. Ε, το άλλο θέμα που τονίζω είναι τα φορολογικά κίνητρα πρέπει να, δεν μπορούμε να δώσουμε ένα συγκεκριμένη εντολή για φορολογικά κίνητρα λόγω των αρμοδιότητων που δεν έχουμε στη φορολογική πολιτική, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε, πρέπει να γίνουν φορολογικές διευκολύνσεις με κρατικές εγγυήσεις, με άλλους τρόπους, ούτως ώστε να αποκτήσουν μια ελκυστικότητα ε, τα σχήματα αυτά. Ε, επίσης πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαστούν οι τράπεζες είναι δύσκολο στι τράπεζε στι συνθήκε που ε, σήμερα έχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα να πούμε ότι θα επενδύσουν σε μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα σχήματα. Πρέπει να δούμε όμω πώ και οι τράπεζε θα το αγκαλιάσουν για να την προσέλκυση των πελατών τους. Ε, επίσης οι περιφερειακές και εθνικές αρχές. Τα σχήματα αυτά, τα ΕΛΤΙΦ, είναι ιδιαίτερα συνδυασμένα με ε, έργα κοινωνικού χαρακτήρα, ε, περιφερειακής ανάπτυξης και πρέπει να δούμε πώς και οι περιφέρειες αυτές θα το ενισχύσουν. Πιστεύω ότι πρέπει να συνδεθούν και με τα project bonds. Δεν μπορώ να πω με τα διαφορετικά ταμεία, διότι τα διαφορετικά ταμεία πρέπει να αποτελούν κάτι πολύ ξεχωριστό, ασφαλές, συγκεκριμένο, αλλά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, με, το, με τα προγράμματα υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ευρύτερα ευρωπαϊκά σχέδια. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια διασύνδεση και ενθάρρυνση από αυτή την πλευρά. Το άλλο θέμα που θέλω να πω είναι τα, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα αξιδοτικά ταμεία που είναι οι κατεξοχήν επενδυτές αυτά. Τα ταμεία πρέπει να δούμε πώς ε, θα διευκολυνθούν από, την, ε, από τις ε, δεσμεύσεις που έχουν ως προς την επάρκεια, από την οδηγία Solvency 2. Πρέπει να δούμε πώς δεν θα ρηψοκινδυνεύουμε την ασφάλειά τους, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να διευκολυνθούν να επενδύσουν, γιατί είναι οι ενδυνάμοι επενδυτές. τονίζω και το σημαντικό ρόλο που έχει ο διαχειριστής, την διευκόλυνση στην ε, αδειοδότηση. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τη ζωή δύσκολη τη στιγμή που το Ταμείο αυτό ε, ε, είναι ένα κομμάτι όλης της ρύθμισης των εναλλακτικών αγορών. Και επίσης ήθελα να τονίζω ότι πρέπει να υπάρχουν και λιγότεροι περιορισμοί όσον αφορά την υποθήκευση των περιουσιακών στα, στοιχείων αυτών των ταμείων. Σε γενικές γραμμές είναι αυτές οι τροποποιήσεις που φέρνω και θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη των σκιωδών και των άλλων εισηγητών και των άλλων μελών της Επιτροπής μας για να συμβάλλουμε σε κάτι ελκυστικό, ασφαλές και αποτελεσματικό ως σχήμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κράτσα από πλευράς των σοσιαλιστών. Ε, έχει το λόγο ο κύριος Χαντράουι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Τα LTF μπορεί να είναι χρήσιμα. Χρειαζόμαστε ένα μέσο το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα να λύσουμε κονδύλια και τα οποία θα επενδυθούν σε επιχειρήσεις και έργα μακροπρόθεσμα ειδικά τη στιγμή κατά την οποία ο τραπεζικός δανεισμός για τέτοια έργα δεν είναι τόσο εύκολος. Οπότε, επί της αρχής είμαστε θετικοί, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα πρακτικά για αυτό το ευρωπαϊκό διαβατήριο, κατά πόσον είναι εφικτό και ασφαλές. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι νομίζω να απευθύνονται αυτά τα προϊόντα και σε θεσμικούς ε, επενδυτές και σε μικροεπενδυτές. Ε, βεβαίως οι μικροεπενδυτές δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι θα δεσμεύσουν τα λεφτά τους για 15 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι πως η Κομισιόν στην πρότασή της ε, ορίζει κάποια πράγματα για το πώς πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους οι μικροεπενδυτές και θεωρώ πως οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει μια κάποια ευελιξία χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει πως θα υπάρχει κίνδυνος για την ίδια τη χρηματοδότηση των έργων. Οπότε με έκανε τη διάκριση μεταξύ μικροεπενδυτών και επαγγελματιών επενδυτών η συγγήτρια. Οπότε έτσι νομίζω απαντάμε στο ερώτημα του κλάδου. Αλλά βεβαίως παραμένει το ερώτημα για το πώς δεν θα διακινδυνεύσει όπως είπα όλη η χρηματοδότηση και ίσως θα ήταν ενδιαφέρον η Κομισιό να μας πει πόσο σημαντικό είναι το θέμα των ιδιωτών επενδυτών ε, και τη συμμετοχή τους είναι δηλαδή κάτι το οριακό ή θεωρούμε πως θα είναι σημαντικό κομμάτι της ε, χρηματοδότησης. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με την πιθανή πρόορη αποχώρηση των ε, ιδιωτών ε, επενδυτών. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τη συμμετοχή τους σε ένα 10-15% του συνολικού έργου. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Δεύτερον, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που θα επενδύουν αυτά τα ταμεία. Μιλήσατε για ε, υποδομές μεγάλης ποιότητας, δρόμους, ε, πιθανώς φυλακές, ε, κοινωνική στέγη, αλλά το, από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες δεν ξέρω δηλαδή αν μπορούσαμε να επεκταθούμε παραπέρα χωρίς ε, κινδύνους. Συμφωνώ με την εισηγήτρια για τις μη εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ε, πιθανούς ε, επενδυτές. Τρίτον, η πρόταση λέει πως θα πρέπει να μπορούν να αγοράζονται και να πολλούνται στη δευτερογενή αγορά μερίδια. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό στην ε, πράξη, ποια θα είναι η αξιολόγησή τους, η αποτίμησή τους. Επίσης βεβαίως θα πρέπει να έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, αλλά οπωσδήποτε, αν είναι σε τρίτη χώρα, οπωσδήποτε όχι σε φορολογικό παράδεισο. για Μπορούμε να δούμε εκεί πέρα τι έχει γίνει και στον κανονισμό κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Δύο πραγματάκια ακόμα τώρα. Μας λέει η συγγήτρια πώς μπορεί ο χρόνος ε, να διαφέρει, να είναι μακράς ε, ή μικρότερης ε, διαρκείας, αλλά νομίζω κάποια συμφωνία θα βρεθεί, θα τις δούμε τις λεπτομέρειες. Και τελευταίο, και σημαντικό για την ομάδα μου είναι βεβαίως η διαφάνεια. Οι επενδυτές ε, στα ταμεία αυτά πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και βεβαίως αυτό αφορά και την αμοιβή των διαχειριστών των ταμείων. Αυτά ως κάποιες ε, παρατηρήσεις. Νομίζω λοιπόν πως θα μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε σε μια καλή πρόταση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αλχαντραουή. Για τους ε, φιλελεύθερους ο κύριος ε, Φιλίπ Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Όπω είπα και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που κάναμε πριν από λίγε εβδομάδε, καλωσορίζω την πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί όντω συμμερίζομαι την άποψη Επιτροπή, όπω και πολλοί συνάδελφοι και παίκτε τη αγορά. Υπάρχει ένα χάσμα επενδυτικό το οποίο πρέπει να καλύψουμε ω προ τι υποδομέ μακροπρόθεσμων επενδύσεων και αυτό θα τονώσει την οικονομία μας, ε, αλλά θα δημιουργήσει και βιώσιμη ανάπτυξη και πραγματικά το χρειαζόμαστε. Ε, όπως λέω και στην έκθεσή μου για τις ΜΜΕ, υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από την δανειοδοσία των τραπεζών και πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό και να κατευθυνθούμε προς ε, μια πολύ πιο διαφοροποιημένη ε, ένα πιο διαφοροποιημένο επενδυτικό σχήμα. Ε, θα ήθελα να κάνω και τρία σχόλια ε, πέρα από αυτή τη θετική αρχική αποτίμηση με, στόχο να βελτιωθεί ίσως το κείμενο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί ιονοί επενδυτές ε, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, για διάφορους τομείς της οικονομίας, για την περιουσία και το καθεξής, αλλά βεβαίως σε σχέση με την περίοδο πρώτης κρίσης θέλουν να αποφύγουν και τον κίνδυνο. Ίσως όμως περιορίζονται και από τον νέο κανονισμό και αποτρέπονται από τις επενδύσεις. Ε, μήπως ε, βεβαίως δεν απευθύνω έκκληση να καταργηθεί ο κανονισμός και να απελευθερωθεί η αγορά και πάλι. Απλώς λέω ότι πρέπει να εξετάσουμε τα κολλήματα για την πλήρη ανάπτυξη ε, του νέου συστήματος των ΕΜΕΚ, των Ευρωπαϊκών Μακροπρόθεσμων Επενδυτικών Κεφαλαίων και να εξετάσουμε και μια σειρά από κανονισμούς που είναι σε ισχύ. Πρόσφατα συζητήσαμε ψηφίσαμε ε, τη, την οδηγία LT4 η οποία ε, ε αναρωτιόμαστε εάν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό το όχημα για τους επενδυτές. Ε, η απάντηση είναι όχι κατά τη γνώμη μας. Ε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να το κάνουν και θα αντενδείκνεται κατά τη γνώμη μου. Είτε θα διαχωρίσουμε σε δύο τμήματα την οδηγία, σε ένα μέρος θα έχουμε τους θεσμικούς επενδυτές με πολύ πολύ αυστηρές ε, διατάξεις ε, και το άλλο μέρος ε, θα αφορά στους ιδιώτες επενδυτές και θα ισχύουν διαφορετικοί όροι. Αυτή είναι η μία λύση. Τώρα, άλλη λύση είναι να επιτρέψουμε στους ιδιώτες επενδυτές ε, να ε, επενδύσουν ε, στο fund of funds, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε και τις δύο λύσεις. Εγώ είμαι ανοιχτός. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ενιαία λύση για όλους. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στους μικροεπενδυτές, στους μεγαλοεπενδυτές, στους θεσμικούς επενδυτές και τους ιδιώτες επενδυτές. Εξαρτάται από τον κύκλο ζωής, από τα δικαιώματα αποζημίωσης που διακρίνουν διακρατούν ή δεν διακρατούν. Υπάρχουν μια σειρά αποζητήματα που πρέπει να συνυπολογιστούν ε, και ε, ε, θα πρέπει να εξετάσουμε ποια στοιχεία των ενεργητικά θα είναι επιλέξιμα για αυτά τα ταμεία. Θα είναι μόνο μακροπρόθεσμες οι επενδύσεις ή θα έχουμε και εισηγμένες εταιρείε και θα έχουμε μερίδια ε, μετοχές και ούτω καθεξής. Ε, θα συνδυάσουμε τους ε, θεσμικούς επενδυτές με τους ιδιώτες επενδυτέ, Πρέπει να εξετάσουμε την μορφή και τη δομή αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων για να πάρουμε αυτές τις επενδύσεις. Μπορούν να γίνουν κάποιες προσαρμογές. Βλέπω ότι η εισηγήτρια είναι πάρα πολύ ανοιχτή και προτίθεται να λάβει υπόψη αυτές τις προτάσεις. Ξαναλέω, πρέπει να εξετάσουμε το πεδίο, τις διαφορές ανάμεσα στους θεσμικούς και τις ιδιώτες επενδυτέ, αλλά Είμαι και ανοιχτό σε σχέση με αυτά που μας είπε ο Σαΐδ για τις τρίτες χώρες και συναφή ζητήματα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι κανονισμοί θα συνάδουν με όσα έχουν αποφασίσει στο παρελθόν και για να μην υπάρχει απόκληση ανάμεσα στις, στις διάφορους κανονισμούς και να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ανασφάλεια στην αγορά και να χειροτερεύσει η κατάσταση αντί να βελτιωθεί. Ευχαριστούμε και ας ακούσουμε και εν τέλει χρονόμος των Πρασίνων τον κύριο Φιλίπ Ντελάμπρεχτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Έχουμε τρεις σκιώδεις Βέλγους. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι τελικά έχουμε πάρα πολλά διαθέσιμα κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να διοχετευτούν προς επενδύσεις. Πάντως, εν γέννη μπορώ να πω ότι χαιρετίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προφανώς χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Τα είπε πολύ καλά ο Φιλίππ. Ας εξετάσουμε αυτή τη στιγμή κάποια σημεία τα οποία θέλουμε να δούμε με την εισηγήτρια. Την δυνατότητα να μπορούμε να μπορούν τα ταμεία αυτά να επενδύουν και σε εταιρείε. Εμείς λέμε ότι ναι, μπορεί να γίνεται αυτό. Δεν Επιτρέπεται όμως από το επενδυτικό ταμείο ανάληψης κινδύνου να επενδύει στο χρηματιστήριο, ενδεχομένω να μπορεί να προβλέπεται κάτι τέτοιο για φάτε ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά ταμεία, εφόσον μιλάμε για άλλου είδους επένδυση. Δεύτερον, οι επενδυτές, οι ιδιώτες επενδυτές, retail investors, συμφωνώ με τον Φιλίπ, δημιουργούμε εδώ πέρα ένα νέο επενδυτικό ταμείο, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι θεσμικοί επενδυτές. Αν θέλουμε να έχουμε όμως και τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια. Έχουν γίνει σχετικές προτάσεις και ήδη στην υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία έχουμε όλους τους μηχανισμούς προστασίας των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα προβλέπεται για τους ΟΣΕΚΑ, τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητικές Αξίες. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την οδηγία ΟΣΕΚΑ προκειμένου να επιτρέψουμε τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών σε αυτά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά ταμεία. Κατά αυτόν τον τρόπο επιλύεται και το ζήτημα της early redemption της πρόορης αποχώρησης και αποζημίωσης των ε, επενδυτών αυτών. Τώρα, όσον αφορά την ε, αναφορά για την ε, περαιτέρω προσαρμογή των κανόνων φερεγγιότητα 2. Εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Είμαστε πάρα πολύ διαλλακτικοί και ελαστικοί στη φερεγγιότητα 2. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προβλέπετε περαιτέρω ε, υπονόμευση των κανόνων αυτών προκειμένου να προβλέπεται και συμμετοχή στα μακροπρόθεσμα αυτά επενδυτικά ταμεία. Τώρα για τις τρίτες χώρες και τη συμμετοχή τους. Ναι, γιατί όχι. Θα μπορούσαμε να εξάγουμε τα ΕΛΤΙΦ, τα ΕΜΕΚ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση όμως αυτή έχει κυρίως ως στόχο να ενθαρρύνει την μακροπρόθεσμη, τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό λοιπόν να επιμείνουμε στο ζήτημα αυτό να πούμε ότι τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια πρέπει καταρχάς να αφορούν κυρίως τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε και την καλύτερη μετάβαση στον ενεργειακό τομέα. Τώρα, για το αν θα πρέπει ε, να προβλέπετε διαφορετική χρονική περίοδος όσον αφορά τον κύκλο ζωής του Ταμείου αυτού. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε από αυτού πολύ ξεκάθαρους κανόνες κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα σχέδιο προτού ολοκληρωθεί, προτού ε, ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του σχετικού επενδυτικού ταμείου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα γίνει με τα οικονομικά αποτελέσματα σε περίπτωση που ολοκληρωθεί το έργο αυτό εν γέρος. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια ότι ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα project bonds. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ομόλογα από τράπεζες ανάπτυξης όπως ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλες σχετικές τράπεζες. Εκεί που έχουμε όμως κάποιες αμφιβολίες είναι το αν θα μπορούσαν αυτά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά ταμεία αφενός να δανείζονται και για το αν τα δάνεια αυτά θα ανταποκρίνονται τελικά στο χρόνο ζωής αυτού του ταμείου. Θα πρέπει επίσης τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά αυτά ταμεία να έχουν μία ξεκάθαρη ανάλυση των περιουσιακών τους ε, στην Χίον. Δεν ξέρουμε ακριβώς αν θα πρέπει να επιτρέψουμε Γι' αυτό το λόγο στα ταμεία αυτά να επενδύουν σε μετοχές βραχυπρόθεσμα στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει τέτοιες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις μέσω μετοχών να λαμβάνουν χώρα γιατί ουσιαστικά κάτι τέτοιο αντιτίθεται στον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των επενδύσεων αυτών. Πέρα από αυτά συμφωνώ με τα υπόλοιπα στοιχεία της ε, έκθεσης αυτής και νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι συμφωνούν άλλωστε. Ε, la Comisión... συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να προσθέσει κάτι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μα ζητήθηκε να δώσουμε κάποια στοιχεία για το ε, σύνολο των επενδυτών που επενδύουν σε τέτοια ε, ΜΕΚ. Στην αξιολόγηση που κάναμε εξετάσαμε τις αγορές που έχουν ιδιώτες επενδυτές και επενδύσει σε ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Στη Γερμανία έχουμε το 70% των ιδιωτών επενδυτών που έχουν επενδυθεί σε τέτοια ΕΜΕΚ. Ε, στα ταμεία ε, οι ιδιώτες επενδυτές ήταν το 30% στα ιδιωτικά κεφάλαια για την περίοδο 2008 έως 2012 και στο Ηνωμένο Βασίλειο το ίδιο. Τα μερίδια των ιδιωτών αντιστοιχούν σε πολύ μεγάλο ε, ποσοστό. Υπάρχει όρεξη δηλαδή από πλευρά των ιδιωτών ε, επενδυτών για να συμπεριληφθούν στο πεδίο αυτής της πρότασης. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Εν τέλει, ακούμε την εισηγήτρια, την κυρία Κράτσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ επικοδομητική αυτή, αυτή η σύντομη συζήτηση. Όλοι συμφωνούμε ότι έρχονται να καλύψουν ε, ανάγκες στην αγορά και στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Περιμένω και τις τροπολογίες των σκεωδών εισηγητών και των άλλων συναδέλφων για να κάνουμε έτσι το κείμενο συνεκτικό και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστούμε κυρία Κράτσα. Η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες είναι η 3η Δεκεμβρίου στις 16 ή 17 Δεκεμβρίου θα εξετάσουμε τις συμβαστικές και στην ΕΚΟΝ θα ψηφίσουμε την 21η Ιανουαρίου. Δεν έχουμε κάτι υπό τα διάφορα. Λία τη συνεδρία. Ευχαριστώ.